Good morning, Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και στα γαλλικά και στα γερμανικά. Sie alle ganz, ganz herzlich Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους θερμότατα στην πρώτη μας συνεδρίαση το νέο έτους. Τα, η αθρώα προσέλευση των μελών μου επιτρέπει να σας καλωσορίσω όλους ε, θερμότατα για την νέα χρονιά και σας εύχομαι σε όλους και σας και τους ε, επισκέπτες μας ό,τι επιθυμείτε για σας και την οικογένειά σας. Υγεία, ευτυχία, καλή επιτυχία, πολύ τύχη και στη δική μας επιτροπή εύχομαι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την καλή, την αγαστή συνεργασία που έχουμε. Αντιπαραθέσεις θα έχουμε και στο μέλλον, ανήκει στη δημοκρατία αυτό και ε, έντονες αλλά η ευπρέπεια επιβάλλεται και η συνεργασία μας. Έχουμε πολλή δουλειά, πολύ περισσότερο από την Πέρση και θα έχουμε και μεγάλη πίεση ε, χρονική για να διεκπαιρεώσουμε τα θέματά μας. Ελπίζω να βρούμε και το χρόνο που χρειαζόμαστε αλλά και την ουσία των θεμάτων. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, καλή χρονιά σε όλους και καλή δύναμη. Χαίρομαι πάρα πολύ που ε, επαρέκαμψε ο αρχηγός ε, επικεφαλής γραμματείας σχεδόν ε, υγιέστατος, έχει αποκατασταθεί πλήρως, όχι εντελώς μετά το τύχημα, αλλά ε, σας εύχομαι περαστικά το συντομότερο. Αρχίζουμε. Θέλω να σας πω ότι αλλάξαμε τη σειρά των σημείων 3 και 4, δεν ξέρω για ποιο λόγο ακριβώς. αφού υπήρξαν αναγκαιότητες που το επέβαλα και ο κύριο Πυρίλο εκπροσωπεί τον κύριο Ντεάντζελη, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Σίγουρα θα το διεκπαιρεώσει θαυμάσια. Περνάω στο σημείο 2, ανακοινώσει. Τελειώσαμε τρία νέο, που είναι το πρώην 4. Ενιαία αγορά για τι επιχειρήσει. και την ανάπτυξη. Κολλείται ο κύριος Αντζελής, ε, όπως σας είπα. Θα δώσω μέσα στο λόγο στον κύριο Πυρίλο για να μας κάνει την εισαγωγή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλή χρονιά και ευόδες των εργασιών όλων μας. Εγώ <coughs> αντικαθιστώ τον κύριο Άντζελης, ο οποίος για πολιτικούς λόγους είναι απόν και μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω και να παρουσιάσω εγώ την ε, ε, την έκθεσή του η ανταγωνιστική αγορά ενέργειας ήταν ένα από τα κεντρικότερα σημεία του ευρωπαϊκού σχεδιασμού και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τα επόμενα χρόνια. Στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης παρακολουθήσαμε την αγορά η οποία σιγά σιγά ε, άλλαζε μαζί με τον κόσμο που άλλαζε και εκείνος οι εργαζόμενοι, οι ε, επιχειρήσεις ε, αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες έχουν πλέον πληγεί από τις οικονομικές διακυμάνσεις και επομένως έχουμε πλέον μπροστά μας ε, μια νέα πρόκληση έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε εμείς σαν Ευρωπαίοι μια προστιθέμενη αξία απέναντι στους ανταγωνιστές μας από τις άλλες χώρες αλλά και σε σχέση και με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του η έκθεση Μόντι είναι εξαιρετικά σαφής. Ε, καταδεικνύει τις ε, ε, δραστηριότητες εκείνες οι οποίες είναι απαραίτητες έτσι ώστε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τις λοιπές επιχειρήσεις να δημιουργηθούν αυτές οι ευκαιρίες οι οποίες θα δημιουργήσουν μία όσο γίνεται πιο διάφανη διαδικασία όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Ε, η τυποποίηση είναι πάρα πολύ σημαντική, η ανάκαμψη ε, της κατανάλωσης ε, καθώς επίσης και αναθεώρηση της υπηρεσίας των του κανονισμού των υπηρεσιών έτσι ώστε να γίνει πιο καλή η κατάσταση για τις επιχειρήσεις. Δεν είναι δυνατόν οι αρχές της αγοράς όμως να ξεχωριστούν από την ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική. Μία, χρειαζόμαστε επομένως μία μια, μια ενεργειακή πολιτική ε, η οποία ε, θα δημιουργεί σωστούς διαδρόμους ε, για την ενέργεια είτε πρόκειται για παραδοσιακές είτε για νέες μορφές ενέργειας. Ε, ανάπτυξη λοιπόν της εσωτερικής αγοράς ε, η οποία θα αντιπροσωπεύεται από την καινοτομία. Στοιχείο απαραίτητο για την επίτευξη των ε, στόχων της στρατηγικής 2020 που αποτελεί και την πραγματική ρόμη της Ευρώπης, την πραγματική δύναμη της Ευρώπης ο συνάδελφος αναφέρει ε, στην έκθεσή του ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία, μεγαλύτερο συντονισμός, εναρμόνιση της χρήσης ε, του ε, φάσματος του ευρωπαϊκού. Και βεβαίως οτιδήποτε υποθεί στην αίθουσα θα το μεταφέρω πιστά στον συνάδελφο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλει κανείς το λόγο, συνάδελφος, αυτή τη στιγμή. Ερωτήσεις έχετε, διευκρινιστικές ίσως. Ή φτάνει για σήμερα, για μια πρώτη εισαγωγή στη συζήτηση. Να Καλώς λοιπόν. Τώρα δεν είναι και ο άλλος συγητής εδώ. Μπορεί να οφείλεται στην αλλαγή της σειράς ή απλώς σε απουσία τους γενικότερη. Ή επίση μπορεί να οφείλεται στο γεγονό ότι αρχίζουμε σε νέα ακριβώ και οι συνάδελφοι δεν έρχονται. Αλλά θα πρέπει να συνηθίσουμε σε αυτό, αλλιώ δεν θα προκάνουμε. Ε, το πρόβλημα είναι οι απόντε. Ωραία. Διεκπερώνεται και το 3. Χαίρετε. Τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Δεν θα περιμένουμε. Άλλη φορά χάσανε οι συνάδελφοι τη σημαντική του τοποθέτηση. Θα την κάνουν άλλη φορά αφού απουσιάζουν. Και πάμε στο επόμενο θέμα. Ε, για τις προτεραιότητες των ενεργειακών υποδομών. Ο εισηγητής είναι ο κύριος ε, Σώσα Βάγνερ και μόλις τελειώσει τις χαιρετούρε και τις ευχές θα του δώσω το λόγο. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ε, πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να εκμεταλλευτώ και εγώ την ευκαιρία, ε, όπως και εσείς και ο Ιταλός συνάδελφος που μίλησε προηγουμένως, για να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά και ό,τι επιθυμείτε στην Επιτροπή μας. Κοιτάξτε, δείτε, τι ωραία ευκαιρία. Ε, μέχρι και συγκινητική θα έλεγα. Το γεγονός ότι σήμερα συζητούμε για τις προτεραιότητες ενεργειακών υποδομών για το 2020 στην Ευρώπη, διότι θα έχετε διαπιστώσει ότι εορτάζουμε την 60η επέτειο της ε, ΕΚΑΧ που είναι ακριβώς ε, η κοιτίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι 60η επέτειος φέτος, είναι πολύ συγκινητικό αυτό και ο Μονέ ο ίδιος, ο οποίος ε, γύθηκε της οργάνωσης αυτής, είχε επιμείνει πάρα πολύ στη σημασία που είχε η ΕΚΑΧ τότε και θα είχε στη συνέχεια για το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση σήμερα και μας επιτρέπει να έχουμε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα λοιπά και να ασχοληθούμε ε, με μια ενεργειακή προοπτική που δεν έχει πλέον καμία σχέση με την προέλευσή της πριν από 60 χρόνια. Είναι πάρα πολύ φιλόδοξη ε, η προσπάθεια αυτή και το εγχείρημα εξαιρετικά επίκαιρο και εύστοχο. Αυτή η ανακοίνωση λοιπόν και η προσπάθεια τι φιλοδοξία έχει. Να στήσει τη σπονδυλική στήλη της Ευρώπης. Τίποτα παραπάνω αλλά και τίποτα λιγότερο. Και επειδή είναι λοιπόν η σπονδυλική στήλη ή η η κοκαλιά θα πρέπει να πούμε ότι δεν φτάνουμε στη συζήτηση αυτή χωρίς προεργασία. Ε, έχουν προηγηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοβουλίες, εργασίες εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ε, δεν είμαστε σε μηδενική βάση σήμερα. Δεν είμαστε οι πρωτόπλαστοι που θα ε, δημιουργήσουμε ε, τον κόσμο από τον παράδεισο, από το μηδέν, όπως σας είπα. Έχουμε ήδη στις αποσκευές μας πολλές κατακτήσεις, ε, πολλά επιτεύγματα από εκείνους που διαχειρίστηκαν την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από εμά. Είχαμε και πράσινες βίβλους και λευκές βίβλους και κανονισμούς και οδηγίες, αλλά κυρίως διατύπωση μια σειρά βασικών θεμελιωδών αρχών που διέπουν ε, την ευρωπαϊκή νοοτροπία για την ενέργεια. Και αυτό τι σημαίνει. Ολοκλήρωση των εθνικών αγορών, εξασφάλιση του ανεφοδιασμού, ε, οικονομία ενέργειας, αηφορία, εναλλακτικά ε, καύσιμα, καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής, τα περίφημα 320 που ε, έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αύξηση των ανανεώσιμων κατά 20% και στη συνέχεια η εντολή μας απορρέει ε, ούτε λίγο ούτε πολύ από τη συνθήκη της Λισαβόνας παρακαλώ. Ε, αφιερώνει ολόκληρο κεφάλαιο ε, και ολόκληρο άρθρο το 194 η συνθήκη που μας υποχρεώνει να δράσουμε. Ε, να ε, υλοποιούμε όλους αυτούς τους στόχους. Επιπλέον θα πρέπει να βγάλουμε και τα απαραίτητα συμπεράσματα, έτσι, ε, τα καθαρά συμπεράσματα από το τρίτο πακέτο εσωτερική αγορά για την ενέργεια. Οδηγίε και κανονισμοί, θυμίζω, που εγκρίθηκαν πάρα πολύ πρόσφατα, το 2009 μόλι. Έτσι λοιπόν, επαναλαμβάνω, δεν είναι ε, νέο έδαφος εδώ τελείως ε, παρθένο. Έχουμε και παράδοση, έχουμε και ιστορία σημαντική ε, στην ενεργειακή αυτή πολιτική μας. Τώρα μόνο συγκεκριμενοποιούνται αυτά τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας. Ένα δίκτυο λοιπόν έχουμε ενεργειακών υποδομών στην Ευρώπη, τη ραχοκοκαλιά όπως σας είπα και πρόοδο μεγάλη στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, διότι σε τελική ανάλυση ο στόχος μας ποιος είναι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταφέρουμε η Ευρώπη να ομιλεί με μία μόνο φωνή σε αυτά τα προβλήματα και σε αυτά τα ευρωπαϊκά προβλήματα. Για να τα επιτύχουμε όλα αυτά λοιπόν, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά κι εσείς ότι χρειάζονται πάρα πολύ στεναρές πολιτικές δεσμεύσεις και πάρα πολύ γενναίες επενδύσεις. Δεν μπορούμε να λησμονούμε εδώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές εντάσεις ακόμα μεταξύ των κρατών μερών, τεράστια ε, αντικρουόμενα εθνικά συμφέροντα, τεράστιος κατακαιρματισμός ε, των ε, αγορών. Τα γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά αυτά τα εμπόδια για να τα ξεπεράσουμε, για να τα ε, υπερβούμε χρειάζεται αποφασιστικότητα και πολιτική ενέργεια και θέληση. Ε, ahora, tenemos que ponernos como objetivos Άμεση λοιπόν στόχη μας θα πρέπει να είναι η εξή. Προσπαθώ να συνοψίσω. Ελπίζω να το καταφέρω. Πρώτον, θα πρέπει να έχουμε τη γενναιότητα να κατονομάσουμε τις απαραίτητες υποδομές, να πούμε τι χρειαζόμαστε για να έχουμε μια κοινή ενεργειακή πολιτική. Άρα, απαρίθμηση πρώτον. Δεύτερον, να ορίσουμε κριτήρια εδώ από το Κοινοβούλιο για να ορίσουμε ακριβώς εκείνα τα έργα που θα χαρακτηριστούν ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας λοιπόν εδώ και να λάβουμε υπόψη μας πάρα πολύ διαφορετικά και ποικίλα στοιχεία. Και αυτό είναι δική μας δουλειά εδώ ε, τους επόμενους μήνες. Ε, ελλείμματα τις υποδομές, ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών κτλ. Αυτά όλα θα πρέπει να τα συμφωνήσουμε. Ένα τρίτο. Εγγύηση τη εκτέλεσης αυτών των έργων σε ένα αλληλογισμένο χρονικό διάστημα. Να βρούμε ε, φόρμουλες για να λυθεί το επίμαχο ζήτημα και καθόδες ε, της ανάθεσης ε, αδειών, της αδειοδότηση καλύτερα στα διάφορα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωση της δίδει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά από τις εφημερίδες και μόνο ότι το θέμα αυτό είναι κομβικό, βασικότατο σε πάρα πολλές χώρες. Οι προθεσμίες για την εκτέλεση, για την υλοποίηση αυτών των μεγάλων έργων επιμηκύνονται, επιμηκύνονται, διονύζονται πολλές φορές και δεκαετίες ολόκληρες. Γιατί υπάρχουν διαδικασίες νομικές, διοικητικές, δημόσιες για να χορηγούνται άδειε, ε, να εγκρίνονται τα διάφορα έργα κτλ. που εξαρτώνται από διάφορους οργανισμούς, από διάφορες αρχές, εθνικές αρχές, περιφερειακές αρχές, τοπικές, ε, δήμους, κοινότητες, οτά κτλ. Και αυτό τι σημαίνει Καμιά φορά ε, ο πληθυσμό ή κάτι και τη περιοχή ε, αντιστέκονται, αντιτίθεται σε κάποιο έργο και το μπλοκάρουν για χρόνια ολόκληρα. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε κάποιου τρόπου να βγούμε από αυτό. Βεβαίω δεν είναι εύκολο και απλό, γιατί έχουμε προβλήματα και στα 27 κράτη-μέλη με την ομοθεσία τους και όχι μόνο αυτό αλλά στις χώρες που έχουν και ομοσπονδιακή δομή περιφερειακή όπως είναι η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία ίδια Καταλαβαίνετε τι γίνεται με τις αρμοδιότητες των περιφερειών σε αυτά τα θέματα και τις εξουσίες. Είναι βασικό λοιπόν αυτό το θέμα κομβικό και θα πρέπει να μας απασχολήσει. Λοιπόν, τι μας προτείνουν ως απάντηση, προβλήματα και ξανά προβλήματα σε όλη την Ευρώπη ατζέντα με διαδρόμου, οριζοντίω και καθέτος. Ε, θα πρέπει να του ορίσουμε ποιοι είναι αυτοί οι διάδρομοι. Η ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει μια πρόοδο για το ποιοι θα μπορούσαν να είναι. Εκεί θα πρέπει να ασχοληθούμε κι εμείς με αυτό το θέμα και να πούμε Μα αρέσουν, δεν μα αρέσουν, συμφωνούμε, διαφωνούμε, τι παρατηρήσει έχουμε, τι σχόλια στις προτάσεις Ευρωπαϊκή Επιτροπής οι οποίε βασίζονται και τεκμηρώνονται πάρα πολύ καλά από τεχνικά κριτήρια. Βεβαίω και υπάρχουν νομοδοτήσει από ειδικού, αλλά αυτά που λέει ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει σώνει και καλά να τα δεχθεί το Κοινοβούλιο. Ε, και εδώ μπορούμε να εισάγουμε και δικά μα κριτήρια. Γνωρίζοντα πάντα ότι το αποφασιστικό είναι να ε, βρεθεί ένα ορισμό για του διαδρόμου και, και να καθοριστούν. Γιατί έτσι ε, αν δεν υπάρχουν αυτοί οι διάδρομοι, δεν μπορούμε να ορίσουμε ενεργειακή στρατηγική πλέον και υποδομές. Θα πρέπει λοιπόν να μας απασχολήσουν αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να τα δουλέψουμε, να τα σκεφτούμε ε, και να κάνουμε τι προτάσει μας. Σας είπα για τη έγκριση, για τις άδειε ε, και κάτι άλλο. Προτείνει κάποιες ε, περιφερειακέ συνενώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλό μου φαίνεται αυτό γιατί είμαστε πάρα πολλά κράτη. Με γεωγραφικέ διαφορέ πολύ έντονες με την ε, γεωγραφική θέση της κάθε χώρας. Άρα λοιπόν έχουμε συνενώσεις. Ξέρω εγώ, οι χώρες της Βαλτικής π.χ. Ε, θα μπορούσα έτσι να ομαδοποιηθεί ε, ένα σύνολο κρατών κάθε φορά. Και ένα από τα τελευταία κεφάλαια θα είναι η χρηματοδότηση όλων αυτών των έργων. Εδώ λοιπόν Θα πρέπει βεβαίως να καλούνται όλες οι ιδιωτικές εταιρείε που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλες business αυτά και θα πρέπει να υπάρξουν και πηγές βεβαίως δημόσιας ε, χρηματοδότησης. Αυτά. Αυτοί είναι λοιπόν οι βασικοί άξονε. Δουλειά πολύ θα έχουμε, μην ανησυχείτε. Θα ήθελα όμω να τονίσω και κάτι άλλο σημαντικό. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρο εύθραυστη, ευαίσθητη από πλευρά ε, ενεργειακή έτσι και ε, αδύνατη, αδύναμη. Από αυτή λοιπόν την ενεργειακή μας αδυναμία θα πρέπει εμείς να αντλήσουμε την απαραίτητη δύναμη για να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη ε, στιβαρή, ισχυρή από πλευράς ενέργειας και στεναρή, άξια διάδοχο της ε, μεγάλης επινόησης της ΕΚΑΧ που σας επαναλαμβάνω ήταν η κοιτίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόλις οριστούν οι ε, σκιώδεις ηγητές από τις διάφορες πολιτικές ομάδες, είμαι πρόθυμος να συναντηθώ μαζί τους την άλλη εβδομάδα ή την παράλληλη για να ε, αρχίσουμε αυτό το διάλογο. Και εγώ θα είμαι πλέον συντονιστής των προτάσεων που θα μου κάνουν οι συνάδελφοι ε, των διαφόρων άλλων πολιτικών ομάδων. Επιπλέον όμως, πέρα από τη δουλειά των εισηγητών και των σχεδόν, για να προχωρήσει η υπόθεση αυτή, τολμώ να απευθυνθώ στους υπολείπους ε, συναδέλφους βουλευτές και να τους πω ότι είμαι στην απόλυτη ε, διάθεση του καθενός και των σκιωδών για να μου διαβιβάσουν τις ανησυχίες τους τις προτάσεις τους, τα μελήματά τους και τα εθνικά βεβαίως που είναι προφανή καμιά φορά και λογικά και τις σκέψεις τους. Είμαι λοιπόν απολύτως στη διάθεσή σας και με ηλεκτρονικά και στο γραφείο μου, με το τηλέφωνο, ό,τι θέλετε. Και με μεγάλη χαρά να σας απαντώ. Είναι μια προσπάθεια όλων μας, της Επιτροπής μας, πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολύ επίκαιρη. Επαναλαμβάνω τώρα στείλουμε τη σποδηλική στήλη της Ευρώπης και θα πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι για να βρούμε λύσεις. Και ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ σύντομα θα συναντηθώ για να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις στη δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ανακοίνωση που είναι βεβαίως πάρα πολύ σωστή και σοβαρή, αλλά χρειάζεται κάποιες διορθώσεις σε κάποιες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κάρενς. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή επίσης. Θα σας δώσω μια απλή εικόνα. Ένα μεγάλο δάσος Στη μια άκρη του δάσους βρίσκεται μια πόλη, στη μέση του δάσους ένα θαυμάσιο ε, εργαστήρι που φτιάχνει πύληνα πράγματα. Αν δεν υπάρχει δρόμος ή μονοπάτι από το εργαστήρι μέχρι την πόλη, είναι αδύνατον ο κεραμοποιός να φτάσει τα προϊόντα του στην αγορά. Το ίδιο περίπου είναι και η ενεργειακή μας υποδομή. Έχουμε πολλά θαυμάσια εργαστήρια και ρίχνοντας όλο και περισσότερα χρήματα σε νέες τεχνολογίες, ορισμένα από τα εργαστήρια αυτά που ίσως υπερπαράγουν ενέργεια δεν καταφέρουν να διοχετεύσουν εκεί στην πόλη που έλεγα πριν που χρειάζεται. Είναι λοιπόν ατελής η υποδομή μας. Είπε έφραστη τουλάχιστον στα αγγλικά που μετέφρασαν εύθραυστη η αγορά της ενέργειας. Εγώ δεν θα την έλεγα έτσι, αλλά σίγουρα είναι ατελής. Εάν ο στόχος μας, και πρέπει να είναι ο στόχος μας αυτός, είναι μια ενιαία αγορά και αυτή η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι στην ουσία το επόμενο λογικό βήμα για την ολοκλήρωση της ενιαία αυτής αγορά. Τα τελευταία, ε, μάλλον πέρσι, εξετάσαμε τρει άξονε της ενέργεια με την έκθεση του Βιδάλ Κουάδρας, για την ασφάλεια της ε, ενέργειας από το αέριο. Δεύτερο για την αποδοτικότητα της ενέργειας του φίλου Μπένσεν. Επιμείναμε πολύ στην ανάγκη δεσμευτικών στόχων. Αν όμως δεν υπάρχει η υποδομή, πολλά από αυτά που συζητούμε για τη στατηγική της ενέργειας, ακόμα και για την προμήθεια αερίου, δεν έχουν νόημα. Αυτό λοιπόν που βλέπω τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πράγματι το επόμενο λογικό βήμα και ένα βήμα που πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά και να υποστηρίξουμε. Μιλούμε συχνά για την ολοκλήρωση, αλλά τουλάχιστον εγώ θα έλεγα να βάλουμε το επόμενο βήμα, να κάνουμε το επόμενο βήμα, ε, το επόμενο σκέλος αυτής της δομής. πολλά στοιχεία διασύνδεσης των διαφόρων δικτύων δεν έχουν δημιουργηθεί γιατί φαίνονται να μην είναι βιώσιμα τουλάχιστον από, τους, από την πλευρά των επενδυτών. Για παράδειγμα για τη Λιθουανία. Καμία ιδιωτική εταιρεία δεν έχει ε, συμφωνήσει, δεν έχει ε, εκδηλώσει ενδιαφέρον για να κατασκευάσει την απαραίτητη αυτή υποδομή διασύνδεσης μεταξύ δικτύων στη Λιθουανία. Προφανώς διότι δεν τα θεωρούν οικονομικά αποδοτικά. Θα δούμε λοιπόν πώς θα μεταφέρουμε την ενέργεια εκεί στην Ευρώπη όπου χρειάζεται. Έχουμε και άλλα προβλήματα τέτοια interconnector, στοιχείων διασύνδεση, που οικονομικά δεν είναι βιώσιμα. Η λύση της Ευρωπαϊκής Επιτροπή είναι να διοχετεύσει χρήματα ευρωπαϊκά στα έργα αυτά που είναι απαραίτητα για να ε, ε, ολοκληρωθεί η αγορά. Αυτό δεν θα γίνει μόνο του βέβαια. Η ανακοίνωση της Επιτροπής τον ίδιο ακόμη την σημασία της συνεργασίας μεταξύ χωρών μελών. Φαίνεται απόλυτα προφανές αυτό για να μειωθεί και το κόστος. Συνοψίζοντας, τονίζω την υποστήριξή μου για την πρόταση αυτή που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επίση, συμφωνώ με την κατεύθυνση του εισηγητού και νομίζω θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι χωρίς αυτό το επόμενο βήμα η νομοθεσία που επεξεργαστήκαμε πέρσι μπορεί εν τέλει να αποδειχθεί ότι είναι ωραία λόγια αλλά που στερούνται νοήματος. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μαδουρέλ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ πρώτα πρώτα θα ήθελα να τονίσω ότι συμφωνώ με τον συνάδελφο εισηγητή για την έκθεση αυτή. Και σας εύχομαι ότι επιθυμείτε για το νέο έτος 2011. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τον εισηγητή με τον οποίο συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό για την πρώτη αυτή ανταλλαγή απόψεων. Ε, από πλευρά τη ομάδα μου ω και ηγητρία θέλω να κάνω μόνο μερικέ σύντομε παρατηρήσει να σα πω μερικέ σύντομε σκέψει για το θέμα είναι πολύ σημαντικό Κοιτάξτε, χωρί, χωρίς να πάμε πολύ μακριά ιστορικά, τόσο μακριά όπως έκανε ο εισηγητής, θα ήθελα να θυμίσω κι εγώ ότι τα τέσσερα τελευταία χρόνια κάναμε ε, πάρα πολύ μεγάλη νομοθετική προσπάθεια για να εμβαθύνουμε στην εσωτερική ενεργειακή αγορά και να ε, βάλουμε στο ενεργειακό μείγμα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά όπως ε, ακούστηκε ε, θα είναι μάταιες οι προσπάθειές μας αν δεν κάνουμε και ένα άλμα στις υποδομές για τη διασύνδεση των υποδομών. Χρειάζεται ένα δίκτυο που να λειτουργεί ε, σωστά χωρίς ε, εσωτερικές αγγελώσεις και στραγγαλισμό. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τους τρεις πυλώνες ενεργειακής πολιτικής που είναι η ανταγωνιστικότητα, η αηφορία, η βιωσιμότητα και η ασφάλεια του ανεφοθιασμού. Σήμερα λοιπόν όλα αυτά είναι γνωστά από τα πιο ε, λοιπόν ασθενή σημεία ο αδύναμος κρίκος είναι οι διασυνοριακές διασυνδέσεις. Ε, ακριβώς ε, επειδή το 2010 δεν προχωρήσαμε πολύ θα πρέπει να επαναλάβουμε ρητά τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για στόχο 10% διασυνδέσεων που είχε αποφασιστεί στο Ευρωπαϊκό Συμβόλιο της Βαρκελόνης. Κατά την άποψή μας θα πρέπει να δοθεί ίδια συνέχεια και σε αυτό το στόχο όπως και στους άλλους για τα 3.20 ε, για τη μείωση ε, των εκπομπών, για τη βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ανάπτυξη υποδομών που θεωρούνται ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος δεν μπορεί να επαφείται μόνο ε, στην επιθυμία δύο κρατών μελών, να βασίζεται μόνο σε αμυγό ως εμπορικά κριτήρια. Γιατί όπως σας είπα προηγουμένως, ε, είναι πολύ μεγάλα τα ωφέλη όταν είναι σωστές οι διασυνδέσεις στην Ευρώπη. Δεν είναι αμυγός εμπορικά συμφέροντα. Γι' αυτό συμφωνούμε απολύτως και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τον εισηγητή για την ανάγκη επιτάχυνσης τώρα των ε, διαδικασιών ε, διοικητικής έγκρισης και διοδότησης των νέων υποδομών. Και όπως δείχνει η εμπειρία, οι καθυστερήσεις και περνούν και τη δεκαετία καμιά φορά χρειάζεται ε, αυτή η ενιαία αντιμετώπιση σε μία και μόνο διοικητική αρχή, σε μία θηρίδα να απευθύνεται κάποιο για να ε, παίρνει ε, την έγκριση και την άδεια. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε και κάποια προθεσμία, μια καταληκτική ημερομηνία για την εκτέλεση των έργων και να βρεθεί ένας μηχανισμός έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να επεμβαίνει σε περιπτώσεις αδράνειας, ολιγορίας από πλευράς εθνικών αρχών. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν θα πρέπει να απευθύνουμε έκκληση ε, στον οργανισμό ε, ρύθμισης ενέργειας ε, που συνδέει τις ρυθμιστικές αρχές να λάβει αυτό το ρόλο. Η χρηματοδότηση θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές της αγοράς όπως πολύ ωραία εξήγησε ο εισηγητής αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να αυξηθούν και οι κοινωτικοί πόροι που αφιερώνονται σε αυτή την προσπάθεια για να αναπτυχθούν οι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος υποδομές γιατί δεν βρίσκουν χρηματοδότηση. Και μια τελευταία σκέψη για τις ανανεώσιμες που είπαν και οι προλαλήσαντες συνάδελφοι. Η συμπρίπτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα επίπεδα που έχουμε θέσει σημαίνει οπωσδήποτε αναδιάρθρωση του ηλεκτρικού δικτύου στην Ευρώπη με συστήματα εφιούς διαχείρισης. Και επί τόπου ε, θα πρέπει να συνδέονται οι μονάδες παραγωγής ανανεώσιμες ε, ε, πηγές ενέργειας δηλαδή, να συνδέονται με το κεντρικό δίκτυο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να εργαστούμε σε δύο κατευθύνσεις την προστασία δεδομένων και την τυποποίηση ε, των υποδομών. Δεν μπορούν να αισθάνονται ανασφάλεια ε, οι καταναλωτές και αυτό να μπλοκάρει την εγκατάσταση εφιών μετρητών ε, του ηλεκτρικού ρεύματος. Θα πρέπει κάποια στιγμή να έχουμε ένα σούπερ δίκτυο, ένα σούπερ grid όπως λέγεται, που να επιτρέπει ε, την ανάπτυξη ε, και ε, τη συνδυασμένη ενέργεια και τις διασυνδέσεις σε σημεία κόμβους, όπως είναι η σύνδεση Ισπανία, Γαλλία και Ευρώπη ή η σύνδεση της αιωλικής ενέργειας που παράγεται εκτικό ρεύμα στη θάλασσα με την ξηρά. Αυτά. Είμαι στη διάθεση του συγητού και είμαι ότι θα έχουμε πάρα πολύ σημαντική συνεργασία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ζαντώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα εξ αρχής να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Σωσο Βάγνερ γιατί είπε μία σειρά πραγμάτων που εγώ θα ήθελα να αναφέρω και τα θεωρώ σημαντικά για αυτό το ζήτημα. Ε, βεβαίως ε, αναφέρθηκε και στη, στον απαραίτητο συντονισμό και στην απαραίτητη συνέχεια και συνέπεια που θα πρέπει να έχει αυτή η εργασία ε, με τα λοιπά προγράμματα ενέργειας έτσι όπως εντάσσονται στα ενεργειακά σενάρια του 2020 και πέραν. Είναι γεγονός ότι φέτος είναι το 60ο γενέθλιο από την γέννηση της ΕΚΑΧ και είναι γεγονός επίσης ότι η ενεργειακή μας κατάσταση και οι ενεργειακές μας ανάγκες δεν είναι ίδιες με αυτές που είχαμε 60 χρόνια ε, πριν και επομένως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι θα πρέπει να πάρουμε σήμερα αποφάσεις οι οποίες θα μας καλύπτουν και για τα επόμενα 60 χρόνια. Και αυτό από μόνο το καταδεικνύει τη σημασία αυτού του θέματος που μας απασχολεί. Ερώτημα λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να εγγυηθούμε ότι θα υπάρχει συνέπεια, συνέχεια της εργασίας αυτής με όσα έχουμε συζητήσει και ψηφίσει στο Κοινοβούλιο μέχρι τώρα. ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Ε, υπό την ηγεσία ε, Μπένσεν ε, ε εμείς ψηφίσαμε ε, για το 20% της ε, ενεργειακής αυτάρκειας ε, μέχρι το 2020 και ανταυτού βρισκόμαστε από την υποπλευρά Κομισιόν με ένα άλλο ενεργειακό σενάριο που δεν λαμβάνει υπόψη ούτε τον δεσμευτικό ή μη δεσμευτικό χαρακτήρα αυτής της δέσμευσης αλλά λέει ότι δεν είναι δυνατόν να εγκριθεί το σενάριο αυτό δηλαδή το σενάριο το οποίο μας υποβάλλει είναι ένα σενάριο το οποίο λέει ότι δεν θα επιτύχουμε μέχρι το 2020 την αποτελεσματικότητα, την, την κατά 20% ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Αυτό όμως θα πρέπει να αποτελέσει βάση της κοινή μας εργασίας και εγώ προσωπικά θα πρότεινα στον εισηγητή ενδεχομένως να συζητήσει ε, με την αντίστοιχη επιτροπή του Κοινοβουλίου έτσι ώστε να εξακριβώσουν την σοβαρότητα του μοντέλου που αποτέλεσε βάση της μελέτης της Κομισιόν. 20% εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι το 2020 δεν είναι λίγο πράγμα. Ε, είναι στην ουσία σαν να είχε κανείς 15 λαμπούκο. Επίσης και στην ανακοίνωση της Επιτροπής είναι γεγονός ότι λαμβάνονται υπόψη μέχρι το 2020 οι στόχοι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά μετά το 2020 διαπιστώνεται μείωση, ε, σημαντική μάλιστα, των επενδύσεων σε ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επομένως θα πρέπει να δούμε το χρονικό όριο του 2020 σαν ένα σηματοδότη που θα οδηγήσει στο 2050 και να πάμε στο 2050 ελπίζω τουλάχιστον με, το, ε, με ένα μεγάλο μέρος, αν όχι το σύνολο ε, της ηλεκτρικής μας ενέργειας που θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά αυτό θα πρέπει να ε, το επιβεβαιώσουμε το 2020. Επίσης, Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι θα πρέπει να γίνει μια ειλικρινή και αντικειμενική συζήτηση ε, για το θέμα της μεταφοράς του άνθρακα και της ε, αποθήκευσης. Στο έγγραφό της η Επιτροπή προβλέπει ε, πολύ σημαντικές επενδύσεις για την μεταφορά του διοξιδίου του άνθρακος ε, και υπάρχουν και πρόσφατα άρθρα ε, για το σταμάτημα τρένων στην ε, Γερμανία και στον Καναδά. Επομένως δεν είμαστε ακόμα βέβαιοι όσον αφορά την τεχνολογία μεταφοράς και επομένως θα πρέπει να βρούμε λογικούς τρόπους και τεχνολογικά σωστούς έτσι ώστε να εντάξουμε τους τρόπους αυτούς ε, στα πλαίσια της ενεργειακής στρατηγικής ε, στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της ε, και καλύτερη αντιμετώπιση και διαχείριση του διοξιδίου του άνθρακος. Θα πρέπει επίσης να κατηγοριοποιήσουμε τα κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την κατάταξη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων τα, για τα προγράμματα υποδομής, για τα σχέδια μάλλον υποδομής, ε, θα πρέπει η Κομισιόν να είναι πιο σαφής, γιατί έχει μπερδέψει λίγο τα κράτη-μέλη. Ε, γιατί θα πρέπει βεβαίως να υπάρχει συνέχεια, συνέπεια ε, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές προοπτικές, αλλά και όσον αφορά τις ενεργειακές και κλιματικές μας προοπτικές. Αυτά με μεγάλη ευχαρίστηση συνεργάστηκα με τον εισηγητή και ε, χαίρομαι πολύ που καταλήξαμε στα συμπεράσματα αυτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ευχαριστήσω καταρχάς τον κύριο Σώσα Βάκνερ, τον εισηγητή, για την ε, παρουσίασή του για αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχουμε μακρά ιστορία καλών προθέσεων και φιλοδοξιών ε, για τη δημιουργία εσωτερικής αγοράς, για την πρόθεση νέων μορφών ενέργειας ε, και για μια άλλη σειρά, μεγάλη σειρά στόχων, φάσμα στόχων. Φοβούμε όμως έχουμε και 100% περίπου σκορ αποτυχίας στην επίτευξη των καλών στόχων μας. Ε, καλό είναι λοιπόν να στοχεύουμε ψηλά, αλλά ακόμα καλύτερο να είμαστε λογικοί σχετικά με την επίτευξη των στόχων. Δεύτερο που ήθελα να πω. Βλέπω εδώ να υπάρχει ένα μείζον πρόσκομο όσον αφορά την χρηματοδότηση αυτών των ε, σχεδίων, ε, ενεργειακών σχεδίων και προγραμμάτων. Ε, υπάρχει ένα ζήτημα οικονομικής ή μάλλον φορολογικής δημοσιονομικής ορθότητας. Ε, όταν ε, καταρτίζουν τους προϋπολογισμούς τους τα κράτη-μέλη και όταν αναφέρονται ας πούμε στα κριτήρια σύγκλησης και τα σχετικά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πάντα πολύ μεγάλη πίεση ε, στον καθορισμό προτεραιοτήτων ε, και την υποστήριξη σχεδίων. Κυρίως δε όταν μιλάμε ε, για σχέδια τα οποία είτε δεν έχουν είτε δεν φαίνεται να έχουν κάποια εμπορικής μορφής αιτιολόγηση και υπάρχουν ε, κάποια προγράμματα υποδομών τα οποία είναι γεγονός ότι ε, δεν έχουν άμεσα εμπορική αιτιολόγηση αλλά έχουν όμως στρατηγική αιτιολόγηση. Ε, και δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλο περιθώριο είτε ο ευρωπαϊκός είτε ακόμα χειρότερα οι εθνικοί προϋπολογισμοί για να συμπεριλάβουν όλα αυτά τα προγράμματα. Επίσης, με πολύ μεγάλη προσοχή άκουσα τον συνάδελφο που μίλησε προηγουμένως και τις παρατηρήσεις, τους, τις παρατηρήσεις του. Επίσης ότι μέχρι το 2050 ανέφερε ότι ε, ελπίζουμε, ευελπιστούμε ότι η ηλεκτρική ενέργεια θα προέρχεται κυρίως, αν όχι εξ από ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας. Μακάρι, μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο, έστω και αν ε, δεν είναι πολύ πιθανό. Όμως απεικονίζεται με τον, με τον τρόπο αυτό και μάλιστα και ο ίδιος παρατήρησε ότι ενδεχομένως δόθηκε υπερβολικά μεγάλη ευελιξία στα κράτη-μέλη όσον αφορά ε, τις του τους ε, για την ενέργεια και ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, πιο αυστηρή νομοθεσία και κεντρικός έλεγχος. Αυτό ε, ε, είναι μια πολιτική σχολή σκέψης που έρχεται, προέρχεται εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων, των, εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι δύσκολο να εφαρμοστεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενδεχομένως και ακόμα περισσότερο. Δεν είναι και εξαιρετικά πρακτικό και ε, λαμβάνοντα υπόψη και τα όσα είπα προηγουμένω για τη χρηματοδότηση, Προφανώ ένα τέτοιο σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Όσον αφορά τώρα τον συντονισμό το, ε, ε, μέσω αυτού του οργανισμού συντονισμού των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας, είναι γεγονός ότι θα πρέπει να παίξει ε, μεγαλύτερο ρόλο, κυρίως όσον αφορά τα συστήματα μετάδοση και τα μεταβατικά συστήματα. Είναι γεγονός πάντως ότι ο ιδιωτικός τομέας, οι επιχειρήσεις, η βιομηχανία ε, είναι και αυτή η οποία περιμένει να δει βελτίωση ε, της κάλυψης των υποδομών στην ε, Ευρώπη και ευελπιστώ ότι θα βοηθήσουν και μπορούν να βοηθήσουν σίγουρα όσον αφορά τον, τις οικονομικές ελλείψεις σταθερά έχουν καταδείξει και οι ρυθμιστικές αρχές το πρόβλημα ε, το οποίο προκύπτει όσον αφορά την συνένεση για την αδειοδότηση. Αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση στην ολοκλήρωση είτε παλαιών προγραμμάτων ενεργειακών είτε νέων. Και εδώ προκύπτει ένα δίλημα. Θα δώσουμε στις αρχές την δυνατότητα να ξεπεράσουν κατά κάποιο τρόπο την υφιστάμενη νομοθεσία ε, και επομένως ε, να δώσουμε στην τοπική δημοκρατία ας πούμε ε, την δυνατότητα να διαμαρτύρεται κτλ. Ε, ή να πούμε ότι ε, οτιδήποτε γίνει δεν θα γίνει δίπλα στο σπίτι μου. Ξέρετε, ακόμα και για αυτές τις πολύ ωραίες ανεμογεννήτριες, για αυτούς τους πάρα πολύ ωραίους ε, ε, ανεμόμυλους της σύγχρονης εποχής, ε, δημιουργούνται πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Επομένως, χρειάζεται όντως κεντρικός σχεδιασμός αλλά ταυτόχρονα συνεννόηση με την τοπική δημοκρατία και τους εκπροσώπους της, δηλαδή τους ντόπιου, τους κατοίκους των περιοχών. Τέλος. Επανερχόμενος στο αγαπημένο μας θέμα, τις ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας. Τίνω να ε, κλείνω προς την άποψη ότι λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες ε, συνθήκες αναρωτιέμαι εάν κάποια κράτη-μέλη θα αναγκαστούν να αναθεωρήσουν τα συστήματα ή τα, σχέδια στήριξης ή επιδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη το τεράστιο κόστος σε σχέση με την επένδυση σε πιο παραδοσιακές μορφές ενέργειας. Και αυτό θα πρέπει να μην το ξεχνάμε. Ευχαριστώ πολύ. Λινέκ. Ευχαριστώ. Εύχομαι με τη σειρά μου σε όλες και όλους τους συναδέλφους ευτυχισμένη την καινούργια χρονιά. Πρώτα για το κείμενο της Κομισιόν. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι η κατάσταση στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας έχει προβλήματα, υπάρχουν, υπάρχει ανάγκη επενδύσεων και ανάγκη βιωσιμότητας. Εγώ θα πρόσθετα μάλιστα ότι πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση των καταναλωτών και κυρίως των μικρών επιχειρήσεων. Προ τετραετίας είχαμε συζητήσει το τρίτο πακέτο ενέργειας και βάλαμε πολλή δουλειά για να κάνουμε την αγορά να λειτουργήσει καλύτερα με την αποδέσμευση των δικτύων από την κυριότητα, δηλαδή να ανοίξουμε τα μεγάλα μονοπόλια, να μπουν στην αγορά περισσότερα περισσότερα μέρη, περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη, περισσότεροι stakeholders. Επίσης, κάποιος μιλεί χωρίς μικρόφωνο και διακόπτη. Επίσης, για να βελτιώσουμε τις επενδύσεις, σημαντικές άλλωστε για τις εναλλακτικές ενέργειες. Εγώ υποστηρίζω τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί. Βλέπω τώρα σε τούτην εδώ την πρόταση ότι σε ορισμένους τομεί έρχεται σε αντίφαση με τις συζητήσει που κάναμε και τις αποφάσεις που λάβαμε πρώτε άρων ετών και που απηχούνται και στο πακέτο οικονομικής ανάκαμψης και στην έκθεση Μπένσιν που συζητήσαμε προ λίγων ημινών. Τα καινούρια NSOE και NSOG που μόλις άρχισαν να λειτουργούν και που ε, η προσέγγιση που επιλέγουν είναι εκ από τα κάτω, ενώ τούτη εδώ η προσέγγιση που προτείνει η Κομισιόν είναι απολύτως από πάνω προ τα κάτω, θα πρέπει πρώτα να αναλύσουμε τις επιπτώσεις που θα έχει η πρόταση που γίνεται τώρα σε ό,τι αφορά την επικουρικότητα, σε ό,τι αφορά την κυριότητα, σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και τους καταναλωτές. Δεν είμαι απολύτως βεβαία ότι ο Επίτροπος γνωρίζει τα πράγματα καλύτερα από τις αγορές. Βέβαια το Κοινοβούλιο σίγουρα τα γνωρίζει καλύτερα από την αγορά. Να είμαστε όμως πολύ προσεκτικοί ε, στην προσπάθεια αυτή μην ανατρέψουμε την ισορροπία που έχει αποκατασταθεί τα τελευταία χρόνια. Σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση δεν βλέπω οι εταιρείε ενέργειας να είναι από τις πιο ευάλωτες στην Ευρώπη για την ώρα. Είναι όλες στέρεες εταιρείε, τα οικονομικά τους είναι σε καλή κατάσταση και ε, αποκομίζουν σημαντικά κέρδη, ακόμη και πέρσι, μέσα δηλαδή στην ύφεση. Δεν είμαι βεβαία λοιπόν ότι το γεγονός ότι δεν επενδύουν σε υποδομές και η χρήση των παλαιών δικτύων επί τόσο διάστημα συνεπάγεται ότι θα πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη ο φορολογούμενος. Θα πρέπει να δούμε ποιος πληρώνει και γιατί πληρώνει σε αυτή την πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική. Διαβλέπω κίνδυνο δηλαδή παράλληλων κινήσεων, παράλληλου σχεδιασμού και ε, διαβλέπω τον κίνδυνο να μην χρησιμοποιήσουμε σωστά τις δυνάμεις της αγοράς όπως θα έπρεπε δηλαδή. Τέλος, θα συμφωνήσω με τον κύριο Τσίτσεστερ ότι οι ρυθμιστές της ενέργειας θα μπορούσαν να παίξουν σημαντικότερο ρόλο. Καθώς επίσης ο τρόπος κατανομής του κόστους στη βιομηχανία, στις μικρές επιχειρήσεις και στους καταναλωτές, αυτό πρέπει να το εξετάσουμε ταυτόχρονα από τη σκοπιά της ανταγωνιστικότητας βλέπω να υπάρχει ένας παραλληλισμός με τις συζητήσεις που κάναμε για την περιαγωγή, το roaming, σε σχέση δηλαδή με το κόστος που μετακυλίεται στο δίκτυο και στους καταναλωτές από τις εταιρείες. Σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης, όπου η τρέχουσα νομοθεσία μπορεί να έρχεται σε αντίφαση με τον κανονισμό περί Συγχαίρω τον εισηγητή και αναμένω με ενδιαφέρον την ε, συνεργασία μαζί του για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Ο Πρόεδρος. Μίλησαν λοιπόν τώρα όλοι οι σκιώδεις συγητές. Στις 10 αρχίζουν οι ψηφοφορίες. Μου μένουν ακόμη 10 εγγεγραμμένοι. Και το θέμα 5 πρέπει να συζητηθεί επίσης πριν από τις ψηφοφορίες. Με δύο λόγια, η μόνη λύση που βλέπω είναι να δώσω το λόγο σε δύο-τρεις συναδέλφους μετά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά να προχωρήσω στην ψηφοφορία. Μετά την ψηφοφορία πρέπει να εξετάσουμε το θέμα 5, ή δεν θα προλάβουμε. Και δυστυχώς οι υπόλοιποι συνάδελφοι θα πρέπει να λάβουν το λόγο σε κάποια επόμενη συζήτηση. Πρέπει όλοι να κάνουμε μια προσπάθεια να είμαστε συντομότεροι. Δεν μπορούμε να έχουμε τόσο ε, φορτωμένη ημερήσια διάταξη και ταυτόχρονα να μιλούν όλοι τόσο πολύ. Ή αλλιώς θα πρέπει να συνεδριάζουμε καθημερινά. Εγώ ευχαρίστως ό,τι απόφαση επιλέξετε, ναι. Αλλά δυστυχώς τώρα αυτό οδηγεί, η κατάσταση σημερινή δηλαδή, στο ότι ορισμένοι συνάδελφοι δεν θα λάβουν το λόγο και αυτό με λυπεί και με δυσαρεστεί. Νομίζω την επόμενη φορά θα βάλω το χρονόμετρο από την αρχή. Κύριε που ήταν, ο κύριος Γιούκ που ήταν μάλιστα και από την αρχή εδώ, από τις 9 ακριβώς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Θα ευχαριστήσω πρώτα τον εισηγητή για την συζήτηση που έχει ξεκινήσει και που νομίζω ότι βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Άλλωστε η έκθεση κινείται προς σωστή κατεύθυνση. Πρώτη ερώτηση που πρέπει να θέσουμε σε αυτούς είναι τι ρόλο μπορούμε να παίξουμε για τις επενδύσεις στον χώρο της αγοράς ενέργειας. Γιατί δεν αφήνουμε δηλαδή τα πράγματα στα χέρια της αγοράς. Εάν παρέμβουμε, ίσως να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα η αγορά, η ενιαία αγορά δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το επιχείρημα. Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η ολοκλήρωση ενιαία αγορά, τα οποία κατά τη γνώμη μου είναι τρία τα εμπόδια. Πρώτα, τα εθνικά συμφέροντα που προτάσσονται των περιφερειακών. Ύστερα, η διαδικασία αδειοδοτήσεως και τρίτο, η τεράστια ζήτηση για τέτοιες υποδομές. Για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια πρέπει να ληφθούν υπόψη στην έκθεση όλες αυτές οι πτυχές. Πρώτα πρέπει να συζητηθεί μια περιφερειακή προσέγγιση και συντονισμός. Για να δημιουργηθεί μια ενιαία αγορά είναι σημαντικό να λειτουργήσουν διαμεθοριακά έργα και να μην επηρεάζονται από εθνικά συμφέροντα. Επομένως, είναι απαραίτητη η διεθνή συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων παραγωγής ενέργειας, καθώς επίσης και για τον καθορισμό των τιμολογίων. Υπάρχουν ήδη σχετικά παραδείγματα, όπως η συνεργασία των χωρών Βίσεγκραντ, όπου πρόσφατα διασυνδέθηκαν τα δίκτυα Ουγγαρίας-Ρουμανίας στον άξονα βορανότου. Αλλά χρειάζεται περισσότερα τέτοια παραδείγματα. Το δεύτερο εμπόδιο είναι η απλούστευση της διαδικασίας αδειοδοτήσεως. Για μεγάλα έργα είναι απαραίτητο να φύγουν από τη μέση παράλληλα έργα, να υπάρξει το λεγόμενο one-stop shop και το τρίτο τρίτο εμπόδιο είναι οι αιτήσει χρηματοδότησης για έργα υποδομής, είπε σχετικά πριν ο κ. Τίτσεστερ. Μέχρι το 2020 χρειάζονται 200 εκατομμύρια ευρώ για έργα μεταφοράς ενέργειας. Τρία, τρεις επενδύσεις μεγέθους Ναμπούκο ανά έτος. Έχοντας αυτό το μέτρο μπορούμε να κάνουμε τους υπολογισμούς τον έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει αυτόν τον τρόπο υπολογισμού και παλαιότερα. Άρα είναι τεράστια η ανάγκη επενδύσεων που σημαίνει ωστόσο και ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο. Μιλούμε για πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ανάγκη και ιδιωτικών επενδύσεων και νέων χρηματοδοτικών μηχανισμών. Αυτές είναι οι τρεις πτυχές λοιπόν που ήθελα να θέσω υπόψη του εισηγητού. Συνοψίζοντας, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή του εισηγητού στην κέντρο ευρωπαϊκή περιφέρεια. Είδαμε στη διάρκεια της οικονομικής κρίσεως πόσο ιστερεί αυτή η περιοχή και αυτό πρέπει να αντιστραφεί. Θα είναι προς το συμφέρον και των ανθρώπων που κατοικούν εκεί αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να προωθηθεί ο διάδρομος μεταφοράς φυσικού αερίου που βορρά προς νότο και ούτω καθεξής. Ε, κύριε Γιόρνταν Σίσελη, ευχαριστώ. Το θέμα αυτό ε, μας έχει απασχολήσει και στην πολιτική μας ομάδα. Το είπε και ο κύριος Ζαντό είπε τι έχει αποφασιστεί. Εγώ θα ήθελα να σας παραπέμψω σε μια συζήτηση που γίνεται στην Ευρώπη και θα συνεχιστεί και φέτος για τις μειώσεις των αερίων του θερμοκηπίου που θα πρέπει να μειωθούν ε, κατά 20% και πλέον. Αν θέλουμε να είμαστε όμως συνεπείς θα πρέπει να ληφθεί και αυτή η πτυχή και στην παρούσα έκθεση υπόψη. Γιατί υπολόγισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα επιβαρεθούν ιδιαίτερα αυτοί οι τομείς της ενέργειας και δεν θα πρέπει να μειώσουν κατά 20% αλλά κατά 34% ε, τις εκπομπές ε, αερίων θερμοκηπίου ε, δραστηριότητες της ενέργειας. Θα πρέπει οπωσδήποτε να το λάβουμε αυτό υπόψη και στα όσα δηλώνουμε και στα όσα ζητούμε. Η 30% μείωση. Λοιπόν, γι' αυτό περιμένω και στα πλαίσια της παρουσίας και του παρόντος εγγράφου να συζητήσουμε για τα προγράμματα αυτά που θα πρέπει να υλοποιούνται στην Ευρώπη, τα επιπλέον έργα, αν θέλουμε να πάμε στο 30% και όχι στο 20% πλέον. Γιατί χρειάζονται και ιδιαίτερα μέτρα, σαν αυτά που πρότεινε και ο Τσάρλς Τσίσεστερ. Καλές σημειώσεις των εκπομπών, μια καθαρή οικονομία, καθαρή κοινωνία, αλλά θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και θα τα λέει και η έκθεση αυτά. Ο συνάδελφος Μπαλτσίτης. E, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα υπόθηκαν πολλά για την ε, κοινή ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Πολιτικά συμφωνούμε. Οικονομικά στην Ευρώπη χωλένουν τα πράγματα. Είναι πολύ σκληρός ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών. Και ένας από τους λόγους είναι η έλλειψη ακριβώς ενεργειακών υποδομών. Ο συντονιστής περιέγραψε την κατάσταση με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια και έωσε και τη γνώμη του για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήταν όμως ε, χρήσιμο και σημαντικό να μας πει κάτι και για το φυσικό αέριο. Τι γίνεται, ας πούμε, το σύστημα αντιστροφής της ροής του φυσικού αερίου. Αλλιώς δεν θα έχουμε ε, ποτέ ενιαία αγορά ενέργειας. Καταλαβαίνω την άποψη που λέει και συμφωνώ ότι δεν, αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν οι διασυνδέσεις. Ε, γι' αυτό χρειάζεται και κίνητρα για να ε, προσελκύσουμε και ιδιωτικά κεφάλαια και ιδιωτικές επενδύσεις. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και να ποντάρουμε όσο γίνεται στη συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα με επενδύσεις για να ε, μπορέσουν να αποδώσουν και οι υποδομές. Οι οποίες δεν θα πρέπει να εκχωρούνται, να εκμισώνονται υπό το μανδύα της ανοικοδόμησης και της βελτίωσης και της αναβάθμισης και της δημιουργίας νέων ε, υποδομών. Λοιπόν, συνοψίζω και λέγω ότι είναι πάρα πολύ καλό το έγγραφο αυτό, αλλά στο μέλλον θα χρειαστεί μεγαλύτερη συνεργασία και θα υπάρξουν και πολύ καλές προτάσεις. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Θέλω να δώσω σύντομα το λόγο στον κύριο Χίλιπρεχτ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με ενδιαφέρον παρακολούθησα τη συζήτηση. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχηθώ καλή χρονιά με κάθε επιτυχία και ευτυχία. Είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με τον εισηγητή τον κύριο Σόζα Βάγνερ. Χαίρομαι για το όσα είπε. Επειδή δεν έχω χρόνο, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να περιστώ σε τρία σημεία. Πρώτον, επιλογή των έργων και των προτεραιοτήτων. Θα πρέπει να διδαχθούμε από το παρελθόν. Ένα με ένα σφάλμα πριν από πέντε χρόνια στα δύο ευρωπαϊκά δίκτυα Χαθήκαμε στι λεπτομέρειε και σε μικροαντιπαραθέσεις, δηλαδή για να υποστηρίξει το δικό σου έργο θα δεχτείς και το δικό μου. Και καταλήξαμε να έχουμε πάνω από 500 έργα, αλλά καμία προτεραιότητα. Κάποια στιγμή σήμερα πρέπει να ε, φτάσουμε στις προτεραιότητες, γι' αυτό ε, υιοθέτησε την πρόταση αυτή top-down ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. κυρία ΕΚ, αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με την προσέγγιση από κάτω προ τα πάνω του Ένσο ΕΚ είναι συμβατά τα προγράμματα αυτά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά ε, υπάρχει ακριβώς η εγγύηση της ευελιξίας που χρειάζεται. Από πολιτικό επίπεδο πρέπει να οριστούν οι μεγάλες προτεραιότητες για να μπορέσουν πλέον οι εταιρείε να ε, μπουν στις λεπτομέρειες για την υλοποίηση των έργων. Σας παρακαλώ να μην ξαναπέσουμε στο ίδιο σφάλμα με έναν τρόπο πάρα πολύ άκαμπτο ε, να ορίζονται και διευθυντικό ε, όλα τα επιμέρους έργα στις λεπτομέρειες τους. Ας τα αφήσουμε αυτό στις εταιρείες που τα εκτελούν. Και ένα δεύτερο είναι οι διαδικασίες έγκρισης και διοδότησης. Όλοι ε, έχουμε κάποιο πρόβλημα με αυτό. Κανείς δεν είναι ικανοποιημένο με τη διάρκεια τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει να συντομευθούν. Αυτό δεν σημαίνει όμω κύριε Τσίστερο, ότι θέλουμε να περιορίσουμε τα δικαιώματα των πολιτών ή τι μελέτε περιβαλλοντικού αντικτύπου να περιορίσουμε. Γι' αυτό Ακούσαμε και αυτά που λένε οι συνάδελφοι από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος ότι ε, ο ε, τράγος για τις καθυστερήσει είναι οι μελέτε περιβαλλοντικού αντικτύπου. Όχι. Μπορούμε να ορίσουμε ένα ε, όριο πενταετία για την απόφαση και μετά από πέντε χρόνια να λαμβάνεται μια απόφαση έστω και αρνητική αντί να εκκρεμεί ένα έργο 15 και 20 χρόνια και να μην ξέρουμε αν μπορεί ή αν πρέπει να υλοποιηθεί. Πιο σύντομε λοιπόν διαδικασίε, με σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών, αλλά να έχουμε και το θάρρο κάποια στιγμή να αποφασίζουμε. Και εδώ η ευθύνη αυτή ε, ε, βαραίνει εκείνου που έχουν την αρμοδιότητα να εγκρίνουν αυτά τα έργα και προσπαθούν να αποποιηθούν την ευθύνη τους αυτή να ε, ξεγλιστρήσουν, δεν λένε ούτε ναι ούτε όχι. Κάποια στιγμή πρέπει ε, να ε, συντομευθούν οι διαδικασίες, να γίνουν πιο αυστηρές χωρίς ε, να περιορίζονται τα δικαιώματα. Και το τρίτο είναι αυτό το πολύπαθο θέμα της χρηματοδότησης και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι σαφές ότι το μεγαλύτερο τμήμα της χρηματοδότηση θα πρέπει να το απομιστεί και να το αναλάβει ο ιδιωτικός τομέας. Δεν διαφωνούμε και εκεί ακριβώς οι ρυθμιστικές αρχές ενέργειας και οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των τιμών. Ε, στο παρελθόν το πρόβλημα ήταν στο λεγόμενο asset setting, δηλαδή περιορίζανε τόσο πολύ ε, το κόστος γιατί δεν ήθελαν ε, οι ρυθμιστικές αρχές να επιβαρύνουν ε, τους τελικούς καταναλωτές στα τιμολόγια. Άρα όμως και οι ενεργειακές επιχειρήσεις περιόρισαν το ενεργητικό τους, περιόρισαν τις επενδύσεις τους γιατί δεν ήταν αυτές αποδοτικές. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν τα ε, σημαντικά κίνητρα για την οικονομία, για την ιδιωτική οικονομία, χωρίς να επιβαρύνεται ο τελικός καταναλωτής υπερβολικά. Αυτό είναι δύσκολο στοίχημα. συμπληγάδε συμπληγάδες, σκύλα και χάριβδη, αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και τέλος, ε, παραμένει και ε, κάποιος χώρος ε, που δεν ενδιαφέρονται οι επιχειρήσεις, έστω και αν έχουν κίνητρα, να επενδύσουν. Ας πούμε σε παραμεθόριες περιοχές διασυνοριακές, αλλά έχουμε καλή εμπειρία με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανοικοδόμησης, που επιταχύναμε ουσιαστικά 15 προγράμματα. Λοιπόν, έχουμε μια ε, περιοχή, ένα υπόλοιπο που μπορεί και πρέπει να δραστηριοποιηθεί και ο δημόσιος τομέας έτσι ώστε να υλοποιούνται ταχύτερα έργα που δεν ενδιαφέρουν τον ιδιωτικό τομέα. Δεν ξέρω με ποια μέτρα και ποιες μεθόδους μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Ε, υπάρχουν ίσως ομόλογα, σδίτες, συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, άμεσες ε, επιδοτήσεις δεν είναι άσπρο μαύρο, χρειάζεται ένα μείγμα και στη χρηματοδότηση. Θα είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση, είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε μαζί στο μέλλον. Κατά τη διάρκεια του έτους 2011 θα βγάλει τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλουμε να ακούσουμε και να λάβουμε υπόψη και τις δικές σας εμπειρίες από την έκθεσή σας όταν θα κάνουμε τις συγκεκριμένες προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ καλή συνεργασία και πάλι. Η κυρία Ερτσόκ, είναι και άλλοι που θέλουν να λάβουν το λόγο για διαδικαστικά. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Λυπούμε λοιπόν, που ζητώ το λόγο. Είναι όμως από τι πιο σημαντικές συζητήσει και λαμβάνοντας υπόψη ότι στι 4 Φεβρουαρίου το Συμβούλιο θα διεξαγάγει συζήτηση σε επίπεδο πρωθυπουργών. Νομίζω θα ήταν πολύ σωστό η Επιτροπή μας πρώτον να μπορέσει να δώσει το λόγο σε όλους όσοι επιθυμούν να μιλήσουν για το θέμα και δεύτερο να βρεθεί τρόπος να <clears throat> σταλεί η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής, της, ε, η γνώμη αυτή της, ε, αυτής της Επιτροπής μας γραπτός στους πρωθυπουργούς που θα συνεδριάσουν στην Ουγγαρία. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Υποθέτω ότι ο κατάλογος των 8 ομιλητών που δεν θα λάβουν το λόγο θα μιλήσουν την άλλη φορά. Και θα έχω εγώ ως πρώτος το λόγο τότε. Απάντηση του Πρόεδρου. Ναι, σαφώς. Ζαντώ. Ναι, Πρόεδρε. Ε, εγώ εγκάλεσα την Επιτροπή σχετικά με, τα, με το μοντέλο που αναφέρει στην ανακοίνωσή της. Ξέρουμε ότι σύμφωνα με το μοντέλο αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη κανένα πρότυπο όσον αφορά την ε, περίοδο μετά το 2020 και επομένως δεν καταλαβαίνω, δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα σε αυτά που γράφει στην ανακοίνωσή της Επιτροπή και σε αυτά που ψηφίζουμε εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο. Χίλμπρεχτ, αν είναι δυνατόν, απαντήστε μας γραπτός. Είναι, είναι θέμα σημαντικό, κεντρική σημασία μάλιστα, που δεν θα έπρεπε να το αφήσουμε ε, ε, ασυζήτητο. Και εγώ το έχω προσέξει αυτό. Καλώς. Σημειώνουμε τα ονόματα των συναδέλφων που δεν μπόρεσαν να λάβουν το λόγο τώρα και εφόσον είναι παρόντες την επόμενη φορά θα τον λάβουν. Ερχόμαστε τώρα στην ε, ψηφοφορία στο θέμα υπαριθμούν 6 πρώτα είναι το θέμα του κυρίου Μπέλετ ελπίζω ότι λειτουργεί το μηχάνημα ψήφι υπέρ της ε, τροπολογίας 21 παρακαλώ σηκώστε το χέρι σας Κατά. Απορρίπτεται. Α, θέλετε επαλήθευση. Καλώς. Το 21 λοιπόν. Επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Μια στιγμή παρακαλώ. Okay. Ναι. Συνεχί... Ε, ε, το επαναλαμβάνουμε, το επαναλαμβάνουμε λέει ο Πρόεδρος. Παρακαλώ επαναλαμβάνετε. 21. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ένας δεν έχει κάρτα. Μία ψήφος παραπάνω του ΕΛΚ από τις προβλεπόμενες. Πέρας της ψηφοφορίας. Εσείς είστε υπέρ ή κατά. Εσείς κύριε Γκέβελς. Άρα 26 υπέρ 23 κατά 27 μάλιστα 22 υπέρ κατά αποχές α συγγνώμη λάθος μου δεν είναι απαραίτητο να ψηφιστεί 22 γιατί καταπίπτει 23 και 8 μαζί, μαζί ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. 24, 38, 43 και 49. Όλες μαζί. Ε, ψήφι, υπέρ. Α, μου φαίνεται ότι το παράκανα στις διακοπές και τώρα δεν είδα ότι και αυτές εκπίπτουν. Υπαριθμούν 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 47 τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11 ψήφοι υπέρ μαζί με την προφορική τροπολογία. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 Εκπίπτει αυτή εδώ. Νο, όχι. Α, όχι. Λοιπόν, η ψήφη υπέρ. Και η 14. Και η συμβαστική 2. Και η 19 και η 66. Όλες μαζί. ψήφοι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Μερικές πάλι εκπίπτουν τώρα και πάμε στις 16, 17, 18 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται ορισμένες πάλι εκπίπτουν τώρα ερχόμαστε στην 30 μάλλον στην 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική 4 Α, 67 θέλετε επαλήθευση. Καλά λοιπόν, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Ορίστε λοιπόν, απορρίπτεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Φεύγουν ορισμένες. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική αξία αν δεν κάνω λάθος έτσι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία επί της αιτιολογικής σκέψης 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ 29, 29, όχι 28, 29. Λοιπόν, 29 υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται μάλλον, ένα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Μετά οι υπόλοιπε εκπίπτουν. Η τρία τώρα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται και αυτή. Τέσσερα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Μετά εκπίπτουν, εκπίπτει η 32, 33 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται μαζί τώρα οι 2, οι 5 και η προφορική τροπολογία επί του 10α. Α, α καποιο δεν το εκπίπτει. Α, λοιπόν, μόνο οι 2 και η προφορική. Yeah, five folds. Yeah, F2 floor. But we vote on the overall amendment of Mr. Kirchner. And number two. Yeah, on block the 33. Oh, it's only necessary to... Χρειάζεται μόνο να ψηφίσουμε την ε, προφορική τροπολογία για το 10α υπέρ κατά εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή οι 7 και οι 35 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μετά εκπίπτουν εκπίπτουν υπαριθμόν 9 Κύριε Σιγητά, συμφωνείτε, ναι. ψηφίσουμε την 9 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρας. 45 υπέρ, 4 κατά. Ωραία λοιπόν. Ακόμη ένας παρακαλώ, ο κύριος Γκέπες που δεν έχει κάρτα. Τελική ψηφοφορία. Επαναλαμβάνεται, έτσι δεν είναι για το νομοθετικού περιεχομένου ψήφισμα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Πέρας. Το ίδιο αποτέλεσμα, 45 υπέρ, 4 κατά και ο κ. Γκέμπελς. Ευχαριστούμε και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ερχόμαστε στην επόμενη ψηφοφορία που είναι το Συμβούλιο Συνεργασίας του Φασικού Κόλπου η Αγγέλικα Νίβλε, η συμβαστική 1, ψήφι υπέρ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 3 υπέρ, ως προσθήκη, όχι. Το λόγο έχει ο κύριος Μπιουτικόφερ, παρακαλώ, υπάρχει πρόβλημα. Πρόεδρε, δυστυχώς δύο παρεξηγήσεις. Πολλές είναι οι δύο, λέει ο πρόεδρος. Δεν είχαμε πει ότι είναι προσθήκη αυτό, αλλά αλλαγή κανονική. Και η δεύτερη παρεξήγηση είναι ο λόγος. Αυτή η ομάδα επιρρογνωμόνων Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεργασίας του κόλπου δεν ασχολείται με την πυρηνική ασφάλεια όπως λέει εδώ. Γι' αυτό κάναμε την πρόταση για αλλαγή. Αν όμως δεν γίνει δεκτή ως αλλαγή θα πρέπει οι συνάδελφοι να το καταψηφίσουν. ως προσθήκη εγώ δεν το βλέπω αλλαγή. Η κυρία Νίμπλερ, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα ε, να το προσθέσουμε γιατί η πυρηνική ασφάλεια είναι ένα θέμα το οποίο επίσης θα πρέπει να συζητηθεί στο Συμβούλιο του Κόλπου. Και παρακαλώ την ομάδα μου να καταψηφίσει την τροπολογία αυτή του κυρίου Μπιτικόφερ. Ψηφίζουμε τώρα την τρία. Όχι προσθήκη, αλλαγή. Όχι προσθήκη, αλλαγή είναι τροπολογία κανονική. Τροποποίηση. Τροποποίηση. Λοιπόν, τρία ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τέσσερα. Κατά τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Αποφασίζεται δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 3 δεν την είδα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέ. κατά αποχές απορρίπτεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία And closed. τέσσερις 44 υπέρ 6 αποχές. Συγχαρητήρια κυρία συνάδελφε, κυρία Νίμπλερ. Επόμενο θέμα. Nein, wir haben hier nichts mehr abzustimmen. Α, δεν έχουμε άλλη ψηφοφορία. Πάρα πολύ ωραία. Λαμπρά. Ωραία. Συνεχίζουμε. Επανερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη στο σημείο 5. Σημείο 5. Απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. In... Ο συνάδελφος Μπελέτ έχει ξανά το λόγο. Είναι το δημιουργικό τμήμα της Επιτροπής μας. Ήβο, σειρά σου. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη που θα με ξαναανεχθείτε, θα ξαναπάρω το λόγο. Μιλάμε τώρα για την ε, δημιουργία και για την ε, απελευθέρωση του δυναμικού κτλ. Θα ήθελα όμως πρώτα απ' όλα να πω κάτι για, τις, ε, για αυτές τις βιομηχανίες παραγωγής ε, ε, πολιτισμού. Ε, μιλάμε για τις επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με την τηλεόραση, με το βίντεο, με τα video games, με τα new media, με τα νέα media τα νέα μέσα ε, και επίσης μιλάμε και για το CCI's Culture and Creative Industries. Ε, μιλάμε επίσης για το design, ε, είτε πρόκειται για τη μόδα, design μόδας, είτε πρόκειται για design γραφικό. Μιλάμε επίσης για τον τουρισμό και την χρήση νέων τεχνολογιών, είτε στον τουρισμό είτε καθαρά τους τομείς νέων τεχνολογιών Αναφέρομαι επίσης και στο, στην πράσινη βίβλα της Επιτροπή όπου γίνεται λόγος για το μεγάλο οικονομικό δυναμικό ε, αυτών των τομέων. Πρόκειται για τους πιο δυναμικούς τομείς, ε, δυνάμει τους πιο, πιο δυναμικούς ε, τομείς των, της οικονομίας, γιατί τώρα συμβάλλουν κάθε χρόνο κατά 2,6% στο ΑΕΠ. 5 εκατομμύρια άνθρωποι ασχολούνται στον τομέα αυτό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως μιλάμε στον τομέα αυτό περισσότερο για μικρές, μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σημαντικός ο ρόλος τους λοιπόν, όχι μόνο στον τομέα της τέχνης αλλά και στον ε, βιομηχανικό τομέα. Ε, μιλάμε ε, εδώ για την δημιουργία νέων τεχνικών, νέας αισθητικής, νέων διαδικασιών και διεργασιών. Στην γνωμοδότηση λοιπόν αυτή τη γνωμοδότηση την οποία έχετε ενώπιόν σας ε, αναφερόμαστε στα προβλήματα τα οποία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτές οι επιχειρήσεις ε, της, του, του CCI. Πρώτα απ' όλα γίνεται σαφής αναφορά στην ψηφιακή ε, ατζέντα που είναι μία από τις ε, κυρίαρχες πρωτοβουλίες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γιατί αναφερόμαστε στην ψηφιακή ατζέντα, μα γιατί θέλουμε να οθήσουμε την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα πραγματικά επιγραμμικό περιεχόμενο έτσι ώστε να δουλεύουν οι επιχειρήσεις αυτές σε ένα ασφαλές ε, ψηφιακό περιεχόμενο και βεβαίως, που προϋποθέτει βεβαίως ε, και την απαραίτητη ευρυζωνικότητα. Ε, και πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία είναι εξαιρετικά σημαντικά για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα στο εγγύς μέλλον. Δεύτερον, πρόσβαση στην χρηματοδότηση. Βεβαίως δεν θα επαναλάβω αυτά που επανειλημμένα έχουμε πει και που αναφέρει έκθεση Σόζα Βάλτερ. Μπορεί να είναι διαφορετικός ο κλάδος, αλλά τα προβλήματα παραμένουν ίδια. Πολλές από τις μικρές ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δρούν στον κλάδο ε, του, του, του πολιτισμού, πάσχουν από το σύνδρομο χρόνιας υποχρηματοδότησης και επομένως ε, χρειάζεται απαραίτητα και γρήγορα ε, venture capital, ε, μοίρασμα κινδύνου, ναι, καινοτόμα χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Αυτά τα αναφέρω διεξοδικά στην γνωμοδότηση, δεν υπάρχει λόγος να τα επαναλάβω. Είναι όμως σαφές ότι περιμένουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παίξει τον ρόλο που της αρμόζει γίνεται λόγος για όλες τις ε, δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν αλλά ε, επίσης και για την ανάγκη ξεκλειδώματος των δυνατοτήτων έτσι ώστε να υπάρξουν και διασυνοριακές επαφές. Ε, ε, ε, πρέπει οπωσδήποτε να ενισχύσουμε τον ρόλο αυτών των επιχειρήσεων του κλάδου CCI έτσι ώστε, αλλά θα πρέπει να τους δώσουμε και την δυνατότητα έτσι ώστε να αναπτυχθούν. Ένα από τα πιο σημαντικά σημαντικές απόψεις ε, αυτή της ε, βιομηχανίας και του θέματος που μα απασχολεί είναι βεβαίως η προστασία ε, των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία. για μία ακόμα φορά και το ζήτημα αυτό δεν είναι νέο, το έχουμε συζητήσει το θέμα της προστασίας ε, της πνευματικής ιδιοκτησίας επανειλημμένα μας έχει απασχολήσει στην Επιτροπή μας αλλά βεβαίως και εδώ ε, στο θέμα των, ε, της βιομηχανίας που δημιουργεί πολιτισμό το, το, CCI δηλαδή οπωσδήποτε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και το ζήτημα αυτό μιλάμε για προϊόντα δημιουργικά μιλάμε για δημιουργία νέων επιχειρήσεων, ε, συγγνώμη, νέων υπηρεσιών, αλλά φυσικά ε, μεγάλη ανάγκη υπάρχει για εξισορρόπηση ανάμεσα στα δύο αυτά σκέλη. Ξέρουμε ότι η Επιτροπή δουλεύει για το θέμα αυτό έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ισορροπημένο πλαίσιο ε, για την ορθή διαχείριση των ε, ε, πνευματικών δικαιωμάτων και της προστασίας των, των πνευματικών δικαιωμάτων και την προστασία και του online περιεχομένου. Και σημαντικό επίσης είναι το ζήτημα των αδειών που δεν θα καλύπτουν μονάχα μια συγκεκριμένη εδαφική περιοχή αλλά που θα αφορούν ε, γενικότερα την χρήση των υπηρεσιών. Ε, το θέμα του ΦΠΑ μας απασχολεί επίσης ε, σήμερα στα περισσότερα κράτη-μέλη οι επιχειρήσεις ε, οι οποίες ε, ασχολούνται με τις καινοτόμες δημιουργίες αντιμετωπίζουν ένα πεπαλαιωμένο καθεστώς ΦΠΑ που αφορούσε τα που αφορούσε υπηρεσίες όχι online αλλά παραδοσιακές Ο ΦΠΑ είναι συνήθως 9 ή 21% ενώ για, τις επιγραμμικές, ε, ε, για την επιγραμμική παροχή υπηρεσιών είναι μηδενικός. Θα πρέπει ε, να δούμε λίγο πώς θα βελτιώσουμε το σύστημα του ΦΠΑ. Αυτά ήταν τα κυριότερα σημεία τα οποία ήθελα να υποβάλω στην Επιτροπή προς ε, σκέψη και συζήτηση, αλλά βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη και τις ε, διοικητικές, τους διοικητικούς περιορισμούς ε, των χρωμοδοτήσεων ε, πρέπει να περιορίσουμε λίγο τον ίστρο μας ε, γιατί είναι άλλη αρμόδια καθήλη επιτροπή αλλά ό,τι μας μου πείτε εδώ θα τα μεταφέρω και στον, στους συναδέλφους Επιτροπής Πολιτισμού. Θα ακολουθήσει η κυρία Ντικάτσετ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ καταρχάς τον κύριο Μπελέτ για γνωμοδότησή του είναι πάρα πολύ καλά εστιασμένη. Έχουμε πολύ συχνά την ευκαιρία να συνεργαζόμαστε στην Επιτροπή Πολιτισμού και δεν με εκπλήσει λοιπόν και η σημερινή του επίδοση. Μερικά σχόλια. Η παγκοσμιοποίηση προκάλεσε ριζικό αναπροσανατολισμό της κλασικής βιομηχανίας Δηλαδή από την παραγωγή αγαθών έχουμε περάσει στις υπηρεσίες και στην καινοτομία. Ο κύριος Μπελέτ ε, τις κατονομάζει πολλές, πολλούς κλάδους οικονομίας που έχουν να κάνουν και της βιομηχανίας με τον πολιτισμό και τη δημιουργία. Σε μεγάλο βαθμό η μελλοντική μας ευημερία θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούμε το δυναμικό μας, τα ταλέντα, τη δημιουργικότητα για να προχωρούμε σε καινοτομία. Και είναι απαραίτητο ε, οι θεσμοί και σε τοπικό επίπεδο, σε περιφερειακό, εθνικό εθνικό και ευρωπαϊκό θα πρέπει να δημιουργούν ευνοϊκό κλίμα με κίνητρα για τις ε, δημιουργικές και πολιτιστικές ε, ε, επιχειρήσεις τη βιομηχανία της Ένωσης. Η πρόταση λοιπόν του κυρίου Μπελέτ μου φαίνεται καλή. συμφωνώ ότι αυξάνεται και η οικονομική σημασία αυτών των κλάδων της οικονομίας και της βιομηχανίας και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Πρέπει όμως να σας πω ότι υπάρχουν ε, τεράστιες δυνατότητες συνεργασίας και συνέργειας σε πολλούς άλλους τομείς, όχι αμυγός δημιουργικούς ή πολιτιστικούς και ε, μπορούν να παίξουν τεράστιο ρόλο σε μια ε, οικονομία που να μην ρηπαίνει και να βασίζεται στη γνώση. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στο σημείο 4 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Θα πρέπει βεβαίως να το λαμβάνουμε υπόψη κάθε φορά που αυτό αποτελεί κίνητρο για να δημιουργεί ο κόσμος, να καινοτομεί, να μελετά, να ερευνά. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να υπάρχει και μια ισορροπία έτσι ώστε να υπάρχει και σωστή πρόσβαση του κοινού και των ενδιαφερομένων σε όλες αυτές τις καινοτομίες. Δεν θα πρέπει να το λησμονούμε. Εγώ είμαι η πρώτη υπέρμαχος και ε, της ε, πολιτιστικής ε, οικονομίας και βιομηχανία και του πολιτισμού γενικότερα, αλλά ε, ξέρω όλα αυτά για τον πλούτο, για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αλλά δεν θα πρέπει ποτέ να λησμονούμε ότι έχει και άλλη πτυχή ο πολιτισμός, που είναι η πτυχή της δημιουργία, της ταυτότητας, του πολιτιστικού πλούτου, παιδεία, και νομίζω ότι εκεί είναι μια λεπτή ισορροπία που θα πρέπει να βρούμε μια καλή διατύπωση για να διαφυλάστε η πρόσβαση στον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την παιδεία, ε, βεβαίω ε, πάντα με σεβασμό και προστασία των δικαιωμάτων πραγματικής ιδιοκτησίας του δημιουργού. Αυτά. Θα τα πούμε κύριε Μπελέτ και όπως πάντα θα συνεργαστούμε αγαστά και θα προσθέσουμε αν θέλετε και αν συμφωνείτε κάποιες δικές μας ιδέες. Ευχαριστώ. Ακολουθεί ο κ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες όπως είπε ήδη ο εισηγητής είναι τομέας κλειδί για την ευρωπαϊκή οικονομία. Αν θέλουμε να μιλούμε για μια πραγματική έννοια αγορά του δημιουργικού τομέα πρέπει να την φροντίσουμε. Η πράσινη βίβλος της Επιτροπής εντοπίζει τους τομείς όπου βλέπει δυνατότητα βελτίωσης. Οι απαντήσεις που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διάρκεια της διαβουλεύσεως δείχνουν καθαρά που πρέπει να ρίξει το ιδιαίτερο βάρος η ψηφιακή ατζέντα που σημαίνει ότι πρέπει να διευκολυθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να παραγάγουν περιεχόμενο γιατί θα οδηγήσει και σε περιφερειακή ανάπτυξη και σε ανάπτυξη πέθρου. Πώς μπορούμε να διευκολύνουμε λοιπόν να κάνουμε καλή, ευκολότερη την ζωή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Χρειάζεται ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο να επιτρέπει κινητικότητα, πραγματική κινητικότητα των ε, φορέων. Μείωση επομένως των οικονομικών και δημοσιονομικών και γραφειοκρατικών εμποδίων, αμοιβαία αναγνώριση, προστασία των καταναλωτών, βελτιωμένη προστασία των καταναλωτών, υποστήριξη των καλλιτεχνών, των αυτά και υποστήριξη βέβαια και διασπορά των βέλτιστων πρακτικών χρειαζόμαστε νέα δημιουργία νέων κέντρων υπεροχής και να απελευθερώσουμε το μεγάλο δυναμικό των μικρών και μισών επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ, κύριε Ούλσφορτ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως ε, πρώην υπουργό Πολιτισμού αισθάνομαι ιδιαίτερη δέσμευση για τον τομέα αυτό. Βρίσκω την πρόταση εξαιρετική. Όπως είπε προηγουμένη συνάδελφος, είναι σημαντικό να αποκατασταθεί μια ισορροπία και μια ανταλλαγή με τον τομέα της παιδείας. Είναι επίσης σημαντικό να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα σε αυτά που οφείλουν να πράξουν οι χώρες μέλη με δημόσιες επενδύσεις και τις πρωτοβουλίες ιδιωτικού τομέα. Και εκεί λοιπόν χρειάζεται μια ισορροπία. Δηλαδή θα πρέπει ο δημόσιος προϋπολογισμός να αναλάβει και αυτός τις ευθύνες του απέναντι στους πολιτιστικούς φορείς που λειτουργούν σε αυτό το πλαίσιο. τα διάφορα ερευνητικά ιδρύματα. Θα πρέπει να συνεργαστούν με την ιδιωτική οικονομία. Δεν μπορούμε να ρίξουμε βάρος μοναχά στα δημοσιονομικά και στον ΦΠΑ. Πρέπει και οι χώρες μέλη βέβαια να αναλάβουν κάποια ευθύνη. να δημιουργήσουν ένα θεμελιώδη μηχανισμό χρηματοδοτήσεων. Σας ευχαριστώ. Η Κομισιόν επιθυμεί να λάβει το λόγο. Ο κ. Πάσκουα. Από τις εμπειρίες που είχα ήδη το Υπουργείο Πολιτισμού μας, λέει ε, ένας ευρωβουλευτής, το οποίο το όνομα δυστυχώς δεν βλέπουμε, έχω να πω το εξής, αν θέλουμε πράγματι να υποστηρίξουμε τον πολιτισμό, πρέπει πρωτίστως να προστατευτεί η πνευματική ιδιοκτησία. Και αυτό στο παγκόσμιο επίπεδο. Διότι πάντοτε θα τίθεται το θέμα αυτό. Πάντοτε θα μας απασχολεί η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, των εμπειριών, Άλλωστε αυτά γίνονται και αντικείμενο εμπορίου. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να προστατεύονται τα δικαιώματα αυτά. Άλλη πρόταση, εν προκειμένου, είναι ότι ίσως πρέπει να απαλλαγεί απολύτως φόρου προσθέμενης αξίας ο τομέας αυτός. Όμως η βιομηχανία της ψυχαγωγίας πρέπει να έχει διαφορετική μεταχείριση από τις ε, βιομηχανίες που την υποστηρίζουν. Αφενός είναι θέμα καινοτομίας, αφετέρου είναι η ψυχαγωγία, δηλαδή η δημιουργικότητα από τη, από τη μια μεριά και η βιομηχανία κάθε αυτή, για παράδειγμα η βιομηχανία παραγωγής ε, δίσκων μέσα στα πλαίσια της βιομηχανίας ψυχαγωγίας. Αυτές είναι οι δύο προτάσεις μου. Ευχαριστώ. Merci, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί η Επιτροπή σας ασχολείται με την πράσινη βίλου της Επιτροπής για τις επιχειρήσεις που δημιουργούν πολιτισμό. Γιατί για να απελευθερωθεί το δημιουργικό πολιτιστικό δυναμικό απαιτούνται υπηρεσίες και απαιτείται κινητοποίηση όλων των πολιτικών και όχι μονάχα ε, των πολιτικών που αφορούν τον πολιτισμό. Νομίζω ότι αυτό είναι και το κεντρικό ενδιαφέρον της Πράσινης Βίβλου και βεβαίως και το μεγάλο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η γνωμοδότησή σας. Πρέπει να επιτρέψουμε, να δώσουμε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις ε, να απελευθερώσουν πλήρως το δυναμικό τους. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται συνεργασία και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και ε, η συντονισμένη συνεργασία των Επιτροπών του Κοινοβουλίου σας. Του Κοινοβουλίου σας. Αυτό κατάφερε να κάνει η Πράσινη Βίβλος τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, αναφέρεστε σε μια σειρά προβλημάτων στη γνωμοδότησή σας, τα οποία προβλήματα όμως ανεφέροντο και στις 350 παρεμβάσεις ε, τις οποίες δεχτήκαμε στη διάρκεια της ε, δημόσιας διαβούλευσης. Νομίζω ότι είναι απαραίτητη η απελευθέρωση του δημιουργικού δυναμικού, όπως ακόμα πιο σημαντική και απαραίτητη είναι η προστασία της ε, του περιεχομένου της πνευματικής και πολιτιστικής παραγωγής, καθώς επίσης και η προστασία ε, των ε, δικαιωμάτων πνευματικής ε, ιδιοκτησίας. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία επανήλθαν στη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης. Θέλω επίσης να αναφέρω ότι βεβαίως πρέπει να κινητοποιηθούν οι διάφορες πολιτικές έτσι ώστε να ε, ελευθερωθεί το δυναμικό των ε, καινοτόμων δημιουργικών και πολιτιστικών ε, βιομηχανιών αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε ότι η απελευθέρωση αυτή δεν αφορά μονάχα και δεν εξαρτάται μονάχα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις, τα όργανα της, αλλά και από τις εθνικές αρχές και ακόμα και τις περιφερειακές αρχές. Χρειάζεται συντονισμός λοιπόν όλων των επιπέδων και όλων των δυνάμεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. 18 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι η προθεσμία κατά ε, για να ε, καταλήξουμε. Ε, σημείο 8. Προκλήσει πολιτική και δημοσιονομική πόρη για μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013. Αυτή είναι μια ιστορία που θέλουμε να διεκπαιρεώσουμε με την επιταχυμένη διαδικασία. Τον Ιούνιο αποφάσισε το Κοινοβούλιο να συστήσει μια έκτακτη επιτροπή που να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, επειδή είναι εγκάρσια η φύση της εντολής αυτής ε, χρειάστηκε να συμπεριληφθούν και οι μεμονωμένες επιτροπές. Γι' αυτό και η Σούρε μας παρακάλεσε μέχρι τέλη Ιανουαρίου να κάνουμε γνωμοδότηση. συντονιστές αρχές Δεκεμβρίου στην τελευταία συνεδρίαση αποφάσισαν να κάνουν μια τυπική ε, επίσημη γνωμοδότηση αλλά με την απλοποιημένη διαδικασία ζητήσαμε από τη Γραμματεία να προετοιμάσει μια τέτοια γνωμοδότηση. Την έχουμε στα έγγραφά μας βασίζεται στα διάφορα έγγραφα της Επιτροπής και θέλω να ευχαριστήσω πολύ τη Γραμματεία και θα πρέπει να φέρουμε σε πέρα σε αυτή τη δικασία. Δεν χρειάζεται να σας διηγηθώ αυτά που λέει το έγγραφο για να συντομεύουμε. Είναι θέματα ενεργειακής πολιτικής, βιομηχανικής πολιτικής, πολιτικής έρευνας, ε, πολιτική διαστήματος, κοινωνία της πληροφορίας. Είναι κάποιες κεντρικές ιδέες για σημαντικά θέματα που θα έχουν επιπτώσει στον προπολογισμό. Να πούμε δηλαδή τι μας ενδιαφέρει. Σε αυτά τα θέματα να μην μας ξεχάσει η δημοσιονομική πολιτική η σημασία της ενεργειακής πολιτικής δεν είδαμε τώρα μόλις η συζήτηση για τις υποδομές, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Η σημασία της βιομηχανικής πολιτικής ε, έχει τονιστεί επανειλημμένα σε διάφορες συζητήσει στην ε, έρευνα και την καινοτομία ακριβώς τα επόμενα χρόνια. Θα πρέπει να βρούμε τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους, όχι μόνο τους υφισταμένους, αλλά και ε, περαιτέρω, αν θέλουμε τις δύο πρώτες ερωτήσεις να δώσουμε απαντήσεις θα πρέπει να βάλουμε το χέρι στην τσέπη και για την έρευνα και για την ε, βιομηχανία. Και τέλος, χωρίς αυτό να είναι ίσονο σημασία, το είδαμε και στο διάστημα ότι έχουμε και οικονομικές συνέπειες. Δεν είναι τόσο απλό αυτό το θέμα σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Είναι λοιπόν ε, ουσιαστικότατο αυτό το θέμα της χρηματοδότησης. Τώρα μην κάνουμε συζήτηση αρχής για όλα τα θέματα. Θα σας είμαι μόνο ευγνώμων αν ε, σύντομα τοποθετηθούν οι πολιτικές ομάδες, οι συνάδελφοι και μετά να φροντίσουμε στη διαδικασία να κάνουμε και αλλαγές στο κείμενο εφόσον απολύτως απαραίτητες. Σας παρακαλώ, όχι όλα τα έγγραφα από την αρχή, πολιτικές τοποθετήσεις να επικεντρωθούμε στα ουσιαστικότερα για μας, για τη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Μερσή δηλαδή. Ο συνάδελφος Γκλάντε ζήτησε πρώτο λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, αφού είναι απλουστευμένη η διαδικασία, εγώ δεν θέλω να την περιπλέξω. Θέλω να πω δύο λόγια κάτι για το τελευταίο, την πολιτική του διαστήματο. Επανειλημμένα είπαμε πόσο προβληματικό είναι. Ακόμα δεν βρήκαμε λεφτά για το Γαλιλαίο και το GMES. Ε, μήπως ε, θα πρέπει να έχουμε ξεχωριστή θέση στον προπολογισμό. Στο 12 να ζητήσουμε ξεχωριστή θέση του προπολογισμού για να ενθαρρύνουμε λίγο και να υποστηρίξουμε και τον Επίτροπό μας και τις υπηρεσίες του. Γιατί ε, από ό,τι φαίνεται υπάρχουν εκεί κάποια κολλήματα, χωλένια, να το πω διπλωματικά αυτή η προσπάθεια. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επίσης στις 7 θέλω να το αλλάξετε. Ωραία, κάντε μια σύντομη πρόταση, λέει ο Πρόεδρος. Καλή ιδέα, εφής. Η κυρία Ρίαρ Μαντουρέλ. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Συμφωνώ με την πρόταση για την απλουστευμένη διαδικασία. Θέλω να σας πω όμως, να σας ανακοινώσω ότι έχω κάποιες σημειώσεις. Ε, έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις, κάποιες σκέψεις μου στη δική μας πολιτική ομάδα. Θα, θέλαμε η έκθεση για την οποία σας εγχαίρουμε και καλή είναι να είναι λίγο πιο έντονη, πιο οξία. Δεν είναι πάρα πολύ διεκδικητική. Αν θέλετε θα σας στείλω μερικά γραπτός θέματα που μας ενδιαφέρει ε, από την ομάδα μας να εκφραστούν με τρόπο ίσως πιο έντονο στην έκθεση. Δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καβάλιο. very much, uh, President. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Κατά κάποιο τρόπο σχεδιάζουμε το μέλλον της Ευρώπης και οπωσδήποτε χρειαζόμαστε και έναν καινοτόμο προϋπολογισμό που θα επιτρέψει ε, την αντιμετώπιση αυτών των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, που έχουμε μπροστά μας. Ε, είμαι και σε... Ε, και στην Επιτροπή ΣΟΥΡΕ ε, και εκεί έχουμε συζητήσει το θέμα και είπαμε ότι θα πρέπει ο προϋπολογισμός να είναι ε, πλέον σχεδιασμένο σύμφωνα με την πολιτική μας ατζέντα γιατί ο σημερινός προϋπολογισμός είναι διαφορετικά σχεδιασμένος. Θα πρέπει να σχεδιάσουμε λοιπόν το προϋπολογισμό σύμφωνα και με την ατζέντα 2020 και να γίνεται συγκεκριμένος λόγος στις πρωταρχικές ε, προτεραιότητε. Δεύτερον, ο προπολογισμό θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τι κοινωνικέ προκλήσει και όλα τα άλλα ζητήματα τα οποία ε, ε, ε, σχετίζονται με τα θέματα τα οποία συζητούμε εδώ στην Επιτροπή Ήτρα και τα οποία άμεσα απορρέουν από τις κοινωνικές ανάγκες. Επίσης, στην έκθεσή σας αναφέρεστε και υπογραμμίζετε την ευελιξία του προϋπολογισμού. Εγώ θα προσθέσω και την απλούστευση του προϋπολογισμού τέλος, το τελευταίο κριτήριο το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσει το πρώτο ε, κριτήριο. Θα πρέπει να αποφασίσουμε ποιες είναι οι πολιτικές οι οποίες θα πρέπει να χρηματοδοτούνται και συγκεκριμένο, στο, στο συγκεκριμένο θέμα πολύ μεγάλη σημασία παίζει η προστιθέμενη αξία η οποία θα πρέπει να είναι υπολογισμένη σε ευρωπαϊκό εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ε, η έρευνα, οι υποδομές είναι πολύ σημαντικά στοιχεία και επομένως θα πρέπει να ε, υπογραμμίσουμε, να υπογραμμίζουμε ε, την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των αποφάσεων που παίρνουμε. Αυτά είναι τα κριτήρια τα οποία θα ήθελα να αναφέρω για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λυπούμε για την υπερβολική ταχύτητα ε, που δεν μας δίνει την δυνατότητα σε εμάς τους βουλευτές ε, να ε, ασκήσουμε το δικαίωμα τροπολογίας και επίσης να πω στην Επιτροπή παρακαλώ υπάρχει κάποιο πρόβλημα Α, όχι ε, όσον αφορά τις ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ε, νέα Ευρώπη. Τέσσερις παρατηρήσεις τώρα. Προτείνεται μια ευελιξία του προϋπολογισμού. Είχα αναφερθεί, κύριε Πρόεδρε, μια ιδέα ότι δηλαδή θα πρέπει να προβλέπουμε, να προβλέψουμε ένα τμήμα που δεν θα αφορά την ευελιξία αλλά την αποτελεσματικότητα. Γιατί εγώ πιστεύω ότι σύμφωνα με τον προϋπολογισμό θα πρέπει, ο προϋπολογισμός μάλλον θα πρέπει να ε, επιτρέπει τον ε, τον πολιετή προγραμματισμό των ε, προγραμμάτων. Στο μέσο της παραγράφου 4, μια και πρόκειται για δημόσιο χρήμα, σας προτείνω να υπογραμμίσετε περισσότερο την έρευνα ε, παρά την ε, ε, χρηματοδότηση των ενεργειακών υποδομών γιατί οι περισσότερες ενεργειακές υποδομές υπογραμμίζονται και προωθούνται βάσει των εμπορικών συμφερόντων και των αναγκών της αγοράς. Λέω λοιπόν ότι θα πρέπει να πούμε οι ενεργειακές υποδομές θα πρέπει να δέχονται δημόσιο χρήμα αλλά και να αποσαφηνίσουμε, αλλά καλύτερα να λέμε ακόμα και τα αυτονόητα, ε, όταν τα προγράμματα αυτά δεν χρηματοδοτούνται από την αγορά. Τέλος, επί της ε, παραγράφου που συνδέεται, που αναφέρεται στην έρευνα, ε, αναφέρουμε ότι χρειάζεται το 1% του ΑΕΠ, αλλά η κεντρική ιδέα για το μέλλον, εξ όσων κατάλαβα τουλάχιστον, είναι να κάνουμε την πρόταση να ευρω... εξευρωπαίσουμε περισσότερο την έρευνα χωρίς ε, ε, να ε, αυξήσουμε τις ενεργειακές εισφορές. Δηλαδή να δούμε τι γίνεται στα κράτη-μέλη και να το εξευρωπαίσουμε περισσότερο. Δεν διαφαίνεται σαφώς. Επίσης μετά δεν γίνεται λόγος για το ίτερ και νομίζω ότι αυτό είναι λίγο υποκριτικό. Τέλος, επί της παραγράφου 11 προτείνω να γίνει ε, λόγος για υψηλή ευρυζωνικότητα και όχι για ευρυζωνικότητα απλώς. Δίστασα äh, προς στιγμή, διότι σκεπτόμουν. Βεβαίως έχουμε όλοι το δικαίωμα να υποβάλουμε τροπολογίες. Έτσι έχουμε συμφωνήσει με τους συντονιστές αλλά σε ταχύτερη διαδικασία, δηλαδή οι τροπολογίες να κατατεθούν στα αγγλικά. Αυτή η συμφωνία έγινε μεταξύ των ιστών. Και η προθεσμία δεν έχει ακόμα εγκριθεί βέβαια, αλλά έχουμε πει μέχρι την 3η 18 Ιανουαρίου στις 12. Ασφαλώς και καθένας μπορεί να υποβάλει τροπολογίες. Το μόνο που παρεκάλεσα είναι να περιοριστούμε σε πραγματικά στα, στα κύρια πολιτικά θέματα. Ο κύριος Ρούμπικ. τονίζω ότι υπάρχει και η συζήτηση περί ιδίων πόρων, own resources. Μην λησμονούμε ότι τα έσοδα από την εμπορία εκπομπών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μείωση των ε, διοξιδίων του άνθρακος. Επομένως μπορούμε εδώ να χρησιμοποιήσουμε για τις δικές μας δραστηριότητες τους ίδιους πόρους. Ευχαριστώ. Τούρμες. Πρώτα-πρώτα <clears throat> Καλή χρονιά σε όλες και όλους τους συναδέλφους που ε, δεν ε, έχω ακόμη ε, χαιρετήσει. Θα είναι δύσκολο το εγχείρημα να προχωρήσουμε τόσο γρήγορα και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να καταθέσουμε τροπολογίες. Εγώ στο σύνολό του βρίσκω το κείμενο αρκετά καλό. Υπάρχει κίνδυνος τώρα, εάν αρχίσουμε να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, να φτάσουμε σε 150-200 τροπολογίες και δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε μετά να τις ε, βάλουμε σε ένα ε, ε, πλαίσιο λογικά συνεκτικό. Ποιες νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι οι προθεσμίες και αν από κάποια στιγμή ξαφνικά έχουμε 150 τροπολογίες ποιος θα τις συνοψίσει. Δεν έχουμε ούτε και συζητητές. Αυτό είναι το διαδικαστικό θέμα που θέτω για να γνωρίζω και ως πράσινη, ως ομάδα πρασίνων, ε, τι προσπάθεια θα πρέπει να καταβάλουμε. Απάντηση του Πρόεδρου. Κοιτάξτε, αυτά τα αποφάσισαν οι συντονιστές. Η άλλη ιδέα που ακούστηκε ήταν να αποσταλεί επιστολή. Όμως η επιθυμία των συντονιστών ήταν να ακολουθήσουμε την διαδικασία που σα εξήγησα. Αυτό σημαίνει ότι όλοι ότι σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες και τον γνωστό μας ζήλο υποβολής τέτοιων, ίσως θα πρέπει να δείξουμε κάποια αυτοσυγκράτηση, να σκεφτούμε ποια είναι τα πιο σημαντικά θέματα που θα πρέπει να θέσουμε με τις τροπολογίες για να μην φτάσουμε στις 150 που λέτε και θα προσπαθήσω μετά σε συνεργασία με την γραμματεία να δούμε ε, πώς μπορούμε να τις κάνουμε δέσμες. Αλλιώς θα προχωρήσουμε με το συνήθι τρόπο, δηλαδή με λίστα ψηφοφορίας. Η δε ημερομηνία ε, για την ψηφοφορία είναι ήδη γνωστή, είναι 27η Ιανουαρίου. Και εάν βέβαια είναι πάρα πολλές τροπολογίες, ασφαλώς περιπλέκεται το θέμα. Όμως, εξετάζοντας το θέμα και ε, εξετάζοντας το κείμενο μάλλον και τους στόχους του, νομίζω και ερμηνεύοντας και τις παρεμβάσεις των συναδέλφων μπορούμε να οργανωθούμε αρκετά καλά. Δελκαστήγιο. Εξ ονόματος της ομάδας μου έχουν υποβληθεί κάποιες τροπολογίες, μάλιστα και εγώ ίδια το έχω κάνει και η συνάδελφός μου Καρβάγιο έχει μιλήσει για τις τροπολογίες που κατέθεσε, αλλά είναι σημαντικό ιδίως στα πλαίσια της συζήτησης και αφού έχουμε αποφασίσει να ακολουθήσουμε την διαδικασία που είπαμε ε, σωστό είναι να ε, πριτανεύσει η κοινή λογική. Εμείς έχουμε καταθέσει 8 έως 10 τροπολογίες. Αυτές είναι όλες. Δεν πρόκειται να υποβληθούν περισσότερες, ε, ίσως, ίσως 2-3 περισσότερες, αλλά πάντως δεν θα ξεπεράσουμε κατά πολύ αυτό τον αριθμό. Και όπως είπαμε ήδη, έχουμε ρίξει το ιδιαίτερο βάρος σε ορισμένα ζητήματα και ωραία θα ήταν να τις προσέξετε τις τροπολογίες αυτές. Τροπολογίες είναι στο κάτω-κάτω δεν είναι έγγραφο άλλου χαρακτήρα. Αν λοιπόν η γραμματεία μπορεί μαζί με τον πρόεδρο να εξετάσουν τις τροπολογίες και βέβαια εφόσον κάποιες έχουν το ίδιο περιεχόμενο μπορούν και να συγχωνευτούν. Σας ευχαριστώ για την υπόδειξή σας. Θα παρακαλέσω οι συντονιστές και στις ε, πολιτικές ομάδες να φροντίσουν ήδη να ε, συντονιστούν οι τροπολογίες. Ασφαλώς και ο καθένας έχει δικαίωμα να υποβάλει τροπολογίες, αλλά ίσως μπορεί να γίνει μια προεπιλογή σε συνεργασία με τους συντονιστές και επομένως να είναι ε, κάπως περιορισμένος ο αριθμός αυτών που τελικά θα υποβληθούν. Πλάσκα. Με την συνάδελφό μου εξετάσαμε την έκθεση και έχουμε καταλήξει σε τρεις συμπληρώσεις. Συμφωνούμε σχετικά με τους μακροπρόθεσμους στόχους για την Ένωση μέχρι το έτος 2050 εν ώψη και της οικονομικής κατάστασης καθώς επίσης και την αβεβαιότητα σχετικά με το από πού θα περάσουν οι αγωγοί είναι σημαντικό να ξεχωριστεί η μακροπρόθεσμη προοπτική από την πιο βραχυπρόθεσμη, η μέσοπρόθεσμη. Είναι σωστό λοιπόν να ξεχωριστούν οι οπτικές αυτές. Και στο θέμα που έχουμε υποβάλει για την κοινωνία της πληροφορίας έχουμε πει ότι ενδιάμεσο στόχος θα πρέπει να είναι η, ευρυ, η ζώνη, η ευρυζωνικότητα. Άλλο θέμα είναι το θέμα των πρωτοβουλειών. Γι' αυτό προτείνουμε οι πρωτοβουλίες στη γνωμοδότηση αυτή να ληφθούν υπόψη πρωτοβουλίες που θα είναι σε θέση να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία απασχόλησης τα επόμενα χρόνια. Και σε ό,τι αφορά την πολιτική για το διάστημα και έχοντας εξετάσει τα όσα προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας, διαπιστώσαμε ότι μας ενδιαφέρει να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ενωμένων Πολιτειών, ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη προσπαθειών. Αυτά. Βεβαίως θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες μέχρι τη 18 πρώτου. Ευχαριστώ κυρία Ερτσόκ. Ε, ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Νομίζω ότι αν η Επιτροπή Ήτρε θέλει ε, να, είναι, να έχει επιτυχία, όπως και εσείς ε, σαν εισηγητής ε, να έχετε επιτυχία, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε μια ενωτική θέση. Όσο είμαστε ενωμένοι, έχουμε πιθανότητα να περάσουμε την θέση μας. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να φιλτράρουμε τις τροπολογίες όπως κάναμε και με τον προϋπολογισμό έτσι ώστε να παραμείνουν μονάχα οι τροπολογίες αυτές οι οποίες παρουσιάζουν ενωτικές θέσεις και οι οποίες ε, αγωνίζονται για κοινέ θέσεις, μακροπρόθεσμες κτλ. Θα ήταν χρήσιμο εάν τα κράτη, εάν, συγγνώμη, τα μέλη τα οποία είναι μέλη και της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμών, ο κύριος Σοντή ας πούμε εγώ Συνάδελφος βάλω εάν ε, θα ήταν καλό λέγω να συναντηθούμε έτσι ώστε να δούμε ε, ποια είναι τα κεντρικά στοιχεία τα οποία θέλουμε να προωθήσουμε γιατί διαφορετικά ε, θα αυξάνεται όλο και περισσότερο ο ρυθμός των ανατροπολογιών και θα κατακρεματιστεί η εργασία μας. Ε, και επομένως το σημαντικό είναι να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να περάσουν περίπου κάποια κεφάλαια ή αν θέλουμε να περάσει οπωσδήποτε το 1α που είναι το κεντρικό μας ε, ε, κεφάλαιο. Έχουμε πρόσφατη την εμπειρία του προπολογισμού του 11. Έχουμε ακόμα νοπές τις μνήμες για την ευελιξία. Ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι εύκολο κεφάλαιο, επομένως να είμαστε να ξέρουμε τι μας γίνεται. σας ευχαριστώ. Διευκρινίστηκαν τα διαδικαστικά. Παράκληση προς τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Κάντε μια... Οργανώστε τις προσπάθειες των πολιτικών σας ομάδων. Είναι και λογικό να συνεργαστείτε κατεξοχήν με τα μέλη ε, της ομάδας σας που είναι και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. και κατά τα λοιπά θα τα επεξεργαστεί αυτά που θα υποβάλλεται η γραμματεία ώστε να ε, γίνουν σύνολα. Επαναλαμβάνω 18 Ιανουαρίου 12η μεσημβρινή προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Το επόμενο θέμα είναι το υπαριθμό 9. Ανάλυση επιλογών για την καταπέραν του 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εκτίμηση του κινδύνου διαρροής άνθρακα. Έχουν ξεκαθαριστεί τώρα τα θέματα σύγκρουση αρμοδιοτήτων με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Αρχίζουμε σήμερα τις διαβουλεύσεις μας. Θα δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Γιόρνταν Σίζελη και μετά στους υπολείπους συναδέλφους που θα ζητήσουν το λόγο. Ρωμάνα, να έχετε το λόγο. Ευχαριστώ αγαπητέ Χέρμπερτ. Σωστό είναι αυτό που είπες. Υπήρξαν πολλές διαδικαστικές δυσκολίες όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα σας εξηγήσω λίγο πώς ε, οργανώσαμε τη διαδικασία για το θέμα αυτό και μετά θα σας πω και το ε, περιεχόμενο, θα αναφερθώ στο περιεχόμενο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να αποφάσισε ότι θα έχει στόχο την μείωση του 20% μείωση των επόμενων ρίων του θερμοκηπίου. Ε, ενώ ε, αποφασίστηκε ότι θα δεσμευθούν και οι υπόλοιπες χώρες με ανάλογες δεσμεύσεις. Ε, μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοίμασε ε, ανακοίνωση με δύο παραρτήματα που έκανε πιο συγκεκριμένο το σενάριο, τουλάχιστον για την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τω μεταξύ έλαβαν χώρα οι διαδικασίες και οι διαπραγματεύσεις του Κανκούν αλλάξαμε τον ορισμό μας και είπαμε ότι θα μειώσουμε τις εκπομπές πέραν του 20% όταν θα υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες τι συνέβη στο Κανκούν. Αυτό θα το πούμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης και επομένως δεν πρέπει να αναφερθώ για το Κανκούν. Η Επιτροπή ετοίμασε μια έκθεση στην οποία να αν τις δυνατότητες, ε, τα πλεονεκτήματα και το κόστος ε, της ε, κατά πέραν του 20% μείωσης και έχει ήδη κοινοποιήσει τα έγγραφα αυτά στα παρατήματα των οποίων βρίσκονται πολλές και ενδιαφέρουσες ε, πληροφορίες. Ούτε ε, σε αυτά τα τρία έγγραφα θα αναφερθώ εν λεπτομερία. Απλώς σας, το λέω για να σας εξηγήσω ποια είναι η διαδικασία. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, είναι αρμόδια επί της ουσίας. Αυτό αποφασίστηκε. Και επομένως η ίδια η Επιτροπή Περιβάλλοντος θα ξεκινήσει η έκθεση πρωτοβουλίας. Όμως αρμοδιότητες επί του θέματος έχει και η Επιτροπή Ήτρε και επομένως θα ακολουθήσουμε τα αναφερόμενα στο άρθρο 50 του κανονισμού. Πράγμα που σημαίνει ότι θα ακολουθήσουμε διαδικασία ε, διτής αρμοδιότητας. Δύο επιτροπές που θα έχουν ε, αρμοδιότητες από κοινού και οι οποίες ε, θα πρέπει να αποφασίσουν από κοινού και το χρονοδιάγραμμα. Επίσης η Επιτροπή Περιβάλλοντος χωρίς ψηφοφορία θα πρέπει να αποδεχθεί τις τροπολογίες ήτρε. Ε, Βεβαίω θα έρθουμε σε επαφή και με την ομάδα εργασία η οποία ασχολείται με τα θέματα αυτά στα πλαίσια της ΕΝΒΗ. Ε, οι πρόεδροι θα έρθουν και αυτοί ε, σε επαφή και η ομάδα εργασίας Ήτρε και η ομάδα εργασίας ΕΜΒΗ θα συναντηθούν έτσι ώστε να προετοιμάσουν την ε, τελική μορφή της έκθεσης. Έτσι θα συνεργαστούμε. Υπάρχουν ε, τομείς ε, όμως αποκλειστική αρμοδιότητα για την επιτοπή Ήτρε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περαιτέρω συζήτηση αλλά και για την προετοιμασία της έκθεσής μας. Ε, στις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε, στην αυτάρκεια ενέργειας, στο eco-labeling, στη σήμανση eco, τη ενεργειακή κατάσταση των κτηρίων, τα smart grids ε, και η καινοτομία. Αυτά θα είναι στοιχεία τα οποία θα αφορούν ε, αποκλειστική αρμοδιότητα. Ενώ θα υπάρχουν και τομείς κοινή αρμοδιότητας, ε, προώθηση πράσινης τεχνολογίας, eco-design κτλ. Αυτή είναι η τομείς τους οποίους ε, θα πρέπει να, με τους οποίους θα πρέπει να ασχοληθούμε. Μέθοδος εργασίας τώρα. Πρώτα απ' όλα το χρονοδιάγραμμα. Σήμερα θα κάνω μόνο μία πρόταση χρονοδιαγράμματος, ε, γιατί θα πρέπει να το συζητήσουμε και με τον εισηγητή της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Στην κατάρτιση της ε, πρότασής μου προσπάθησα να λάβω υπόψη ε, και τις υποχρεώσεις της Επιτροπής Ήτρε αλλά ε, και το μέλημα για γρήγορη και αποτελεσματική διαδικασία στο μέτρο του δυνατού φυσικά. Περιμένω ότι θα έχουμε πολλές τροπολογίες, επομένως θα πρέπει να έχουμε και χρόνο έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιες συμβιβαστικές λύσεις. Ξέρετε ότι θα πρέπει ε, να υπάρξει συμφωνία στα πλαίσια της Ήτρε, συμφωνία στα πλαίσια της ΕΜΒΗ και συμφωνία μεταξύ των δύο επιτροπών. 21 Φεβρουαρίου λοιπόν ή μάλλον μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου ε, θα έχουμε ε, τον χρόνο, εγώ δηλαδή θα έχω τον χρόνο να προετοιμάσω την έκθεση. Μετά 14 ή 15 Μαρτίου στη συνεδρίαση Ήτρε θα συζητηθεί η έκθεση. 24 Μαρτίου η προθεσμία υποβολής τροπολογιών, τροπολογίες που θα συζητηθούν στην Επιτροπή 12 και 13 Απριλίου 25-26 Μαΐου θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε στην Επιτροπή Ήτρε. Αυτή είναι η πρόταση χρονοδιαγράμματος που κάνω, που βεβαίως όμως θα πρέπει να τη συζητήσουμε και να τη συμφωνήσουμε και με την ε, Επιτροπή. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος προγραμματίζει και σχετική ε, ακρόαση. Προχθές ε, μου το είπαν. Πρέπει να πω ότι η ακρόαση αυτή μου προκαλεί κάποιο προβληματισμό και κάποια σχόλια. Ε, ή θα πρέπει να είναι κοινή ακρόαση ΕΜΒΙΤΡΕ, θα λάβει χώρα στις 28 Φεβρουαρίου και αν καταφέρουμε να έρθουμε σε συμφωνία με τον εισηγητή της Επιτροπής Περιβάλλοντος ε, τότε θα εγκριθεί το χρονοδιάγραμμα. Εάν όμως δεν, δεν υπάρξει συμφωνία μαζί του προτείνω να οργανώσει η Ήτρε δικιά της ακρόαση γιατί πρόκειται για μια έκθεση και ε, μια απόφαση εξαιρετικά σημαντική. Άρα θα πρέπει να ε, ε, προετοιμάσουμε και εμείς, να προβλέψουμε και εμείς μια ακρόαση. Πράγμα που σημαίνει βεβαίως ότι θα μετακυλιστεί λίγο περισσότερο, λίγο πιο αργότερα το χρονοδιάγραμμά μας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι σήμερα ήδη έχουμε το 20%, έχουμε συμφωνημένο το 20% της μείωσης των εκπομπών αερίων και θέλουμε να προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να ε, δούμε εάν όντως θέλουμε να πάμε πέραν του 20% ή όχι. Θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τον τρόπο και με τον χρόνο που θα γίνει κάτι τέτοιο. Κυρίως όμως θα πρέπει να ασχοληθούμε με τις προϋποθέσεις οι οποίες είναι απαραίτητες ε, για να ε, ξεπεράσουμε το 20% και γιατί πρέπει να ξεπεράσουμε το 20%. Ε, εγώ θα ήθελα να χωρίσω την σκέψη μας σε κάποια κεφάλαια. Πρώτα απ' όλα, τον τομέα της ενέργειας. Το κεφάλαιο αυτό της ενέργειας θα ασχοληθούμε ασχοληθώ με την συμβολή της ενέργειας στη μείωση των εκπομπών αερίων και βεβαίως θα αναφέρουμε και τις προσδοκίες μας όσον αφορά την παραγωγή, ε, όσον αφορά την ενεργειακή αποτελεσματικότητα, όσον αφορά ε, την ενεργειακή αποτελεσματικότητα των ε, κτηρίων, τους έξυπνους μετρητές κτλ. Μετά θα μιλήσουμε οπωσδήποτε και για τις σχέσεις με την βιομηχανία, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αναφορά και στην ε, μεγάλη χρήση ενέργειας, στις ε, εναλλακτικές μορφές ε, ενέργειας και την τομεακή προσέγγιση θα πρέπει να αναφερθεί επίσης. Επόμενο κεφάλαιο. ανταλλαγή εκπομπών, συμβολή της έρευνας, αποσαφήνιση του στόχου της μείωσης. Και ένα άλλο κεφάλαιο, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα αναφέρονται στα προηγούμενα κεφάλαια αλλά εν συνθέσει και οπωσδήποτε λαμβάνοντας υπόψη και τις εξωτερικές συνθήκες ε, δηλαδή όχι μονάχα να βλέπουμε τι θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Εγώ θα, θα προτίθεμαι να υπογραμμίσω ε, την παροχή κινήτρων ε, καθώς επίσης και την χρηματοδότηση γιατί θεωρώ ότι είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά κεφάλαια και εν συνθέσει θα πω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μία ε, θετική πολιτική, μία, μία ενεργητική πολιτική η οποία θα μας οδηγήσει στα αποτελέσματα τα οποία θα επιθυμούσαμε. Αλλά βεβαίως να μην ξεχνούμε και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάκαμψη της οικονομίας και για την ε, ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Συχνά λέγεται ότι λόγω της χρηματοπιστωτικής ε, κρίσης οι δαπάνες οι οποίες ε, αφορούν την επίτευξη των στόχων είναι χαμηλότερες αλλά βεβαίως είναι μικρότερα και τα έσοδα των ε, επιχειρήσεων. Άλλωστε έχει πέσει και η αγοραστική δύναμη των αγοραστών. Άλλωστε πολύ πιο δύσκολα πλέον παίρνει κανείς οποιαδήποτε μορφή δανείου από τις τράπεζες. Επομένως θα πρέπει ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλα τα στοιχεία αυτά όταν έχουμε μπροστά μας έναν τόσο φιλόδοξο στόχο όσο η μείωση των εκπομπών αερίων. Ε, τέλος να σας πω ότι δεν έχω ακόμα συναντήσει τους ε, σκιώδεις Ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα μπορέσω να τους συναντήσω έτσι ώστε να συμφωνήσουμε επί της θέσεως που θα πάρουμε και τους, της με την ΕΜΒΗ. Σας ευχαριστώ πολύ και για την ε, εξαιρετικά λεπτομερή παρουσίαση της διαδικασίας, κάτι το οποίο είναι απολύτως χρήσιμο, γιατί είναι πάρα πολύ περίπλοκη η διαδικασία. Έχω τώρα εννέα εγγεγραμμένους και ούτε καν δέκα λεπτά. Να δούμε λοιπόν. Παράκλησή μου είναι, αν ο καθένας σας μπορεί να τα πει πολύ γρήγορα, πολύ συνοπτικά. Θα βάλω το χρονόμετρο να μιλήσει ο καθένας από ένα λεπτό. Δεν θέλω πάλι οι τελευταίοι να μην λάβουν το λόγο. Αν κάνουμε όλη μια προσπάθεια νομίζω θα προλάβουμε. Άλλωστε πρόκειται για την πρώτη φάση της συζήτησης και κυρίως να ξεκαθαριστεί η διαδικασία. Εκ, η κυρία Εκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την θαυμάσια δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα και που αναμένω να κάνει και μετά. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς οι διάφοροι μηχανισμοί που διαθέτουμε αποδίδουν αποτελέσματα. Μιλούμε <clears throat> για νομοθεσία, για standard setting όπως για την αυτοκινητοβιομηχανία και τέλος για οικονομικά κίνητρα και ε, αντικίνητρα και πώς θα λειτουργήσουν στον τομέα αυτό. Θα είναι ενδιαφέρον νομίζω να συζητήσουμε τις διάφορες μεθόδους που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο νομοθέτης εν προκειμένου. Και συζήτηση επίσης των διαφορών μεταξύ των χωρών μελών. Κάθε χώρα μέλος έχει κάποιο προτιμόμενο θέμα για την εναλλακτική ενέργεια, είτε πρόκειται για την νεολική, είτε πρόκειται για την ηλιακή και ούτω καθεξής. Βλέπουμε τομείς αλλά και περιφέρειες όπου η καθεμιά έχει τη δική της προτίμηση και σπάνια βλέπουμε όλες τις εναλλακτικές ενέργειες μαζί. Έχουμε λοιπόν μια εικόνα της Ευρώπης που δεν είναι όμως απολύτως αληθινή ότι δηλαδή η Ευρώπη τα πάει πολύ καλά, έχει πρώτο πόρο ρόλο. Η Κίνα μέσα σε μια δεκαετία από 0% ποσοστό, μερίδα δηλαδή, μερίδιο μάλλον τη παγκόσμια αγορά στην ολική ενέργεια έχει φτάσει στο 50%. Εξαιρετικά σημαντικό παράδειγμα αυτό για να δούμε οι νέε τεχνολογίε, η καινοτομία στον τομέα αυτό, τι μπορεί να προσφέρει σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας καθώς και την οικονομική ανάπτυξη της Υπήρου. Εν τέλει, για το θέμα της διαρροής διοξιδίου του άνθρακος, τη διαρροή δηλαδή ε, των επιχειρήσεων, ε, το ενδεχόμενο μετακίνησης επιχειρήσεων από την μετεγκαταστάσεως επιχειρήσεων από την Ευρώπη λόγω της αυστηρής νομοθεσίας στο θέμα αυτό, εγώ βλέπω να είναι παρόμοιο το φαινόμενο όταν συζητούμε δηλαδή για την εντό εισαγωγικών διαρροή λόγω ε, του διοξιδίου του άνθρακα, διαρροή επιχειρήσεων στην πραγματικότητα, με αυτήν τη συζήτηση που γίνεται για το κλίμα. Η κατάσταση δεν έχει γίνει τόσο δραματική όσο την είχαν προείπει ορισμένοι εκ των ενδιαφερομένων. Η μέθοδος εργασίας που προτείνει η συγγήτρια είναι καλή Νομίζω θα χρειαστεί κάποιο είδου ακρόαση με εμπειρογνώμονε για να ενημερωθούν οι βουλευτέ για, για τα θέματα αυτά. Και η συζήτηση για το τι έγινε στο Κανκούν, πώς θα προετοιμαστούμε για την επόμενη ε, διάσκεψη στην ε, Νότια Αφρική. Ευχαριστώ. Καστίγιο. Καλά, θα προσπαθήσω να περιοριστώ σε ένα λεπτό. Πρώτα συγχαρητήρια στην εισηγήτρια που έχει συντάξει ένα σχέδιο εργασίας πραγματικά εξαιρετικό και το σχέδιο εκθέσεως διαγράφεται πολύ ενδιαφέρον. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε πρώτα πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση σχετικά με τα συμπεράσματα του Κανκούν, στο φως των οποίων θα μπορούσαμε να προβλέψουμε ίσως μια άλλη προοπτική μια άλλη οπτική αν θέλετε για την έκθεσή μας. Είναι κρίμα που δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Τώρα για την ίδια την έκθεση νομίζω ότι τίθεται δύο θέματα. Πώς θα ξεπεράσουμε το 20% πρώτο. Δεύτερο, τι γίνεται με το ε, περίφημο carbon leakage, δηλαδή με την κατάσταση επιχειρήσεων λόγω ε, αυστηρών αριθμίσεων για το διοξείδιο του ανθάκα. Λοιπόν, τώρα είπαμε πρώτα μείωση του κόστους. Όπως είπε η Ρωμάνα η συγγετριά μας, υπήρξε όντως μείωση των εσόδων των επιχειρήσεων. Αυτό ναι, αν όμως μειώθηκε και το κόστος, τόσο καλύτερο. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Να είμαστε λοιπόν καλύτερα προετοιμασμένοι στον αγώνα κατά αυτού του carbon leakage. Θα πρέπει λοιπόν να εκμεταλλευτούμε τα πλεονεκτήματα που διαθέτουμε. Αυτά για το πρώτο. Υπάρχει μια διαφορά φάσης βέβαια με αυτά που συνέβαιναν προηγουμένω. Για τα υπόλοιπα τώρα, ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει ενδιαφέρουσε προτάσεις, πρόσθετε προτάσει για τους ιδιαίτερα ενεργοβόρους τομείς. Αυτό με ενδιαφέρει. Νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας ένα έγγραφο που έχει ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Τέλος πάντων, όπως και να είναι, ό,τι και να γίνεται στο υπόλοιπο του κόσμου, εμείς πρέπει με κάποιο τρόπο να θέσουμε το θέμα του 30%. Ζαντώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την εισηγήτρια γιατί πιστεύω ότι με ορθότατο τρόπο αναφέρθηκε σε όλα τα στοιχεία ε, τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Όσον αφορά τον, το χρονοδιάγραμμα, άλλωστε αυτό είναι ο στόχος μας, να έχουμε δηλαδή ε, το θέμα στην Ολομέλεια πριν από το Συμβούλιο του Ιουνίου. Επομένως ε, θα πρέπει να πάρουμε απόφαση πριν από την συζήτηση και την απόφαση του Συμβουλίου. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που διέπει το χρονοδιάγραμμα. Επί των διαφόρων σημείων που ανεφέρθησαν. Ένα. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό, το είπε άλλωστε και η συγγήτρια, να έχουμε φιλόδοξο στόχο όσον αφορά ε, την ε, κλιματική αλλαγή, αλλά χωρίς να ξεχνούμε και την ανταγωνιστικότητα. 200 δις ε, δολάρια έχει η Κίνα στο πρόγραμμα ανάκαμψή της. Ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε επίσης, ε, η Νότια Κορέα κρατούν τα ενία. Δυστυχώς η Ευρώπη είναι πιο πίσω. Σύμφωνα με το βαρόμετρο 2010, όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Κίνα και η ΙΠΑ κρατούν τα ενία και για τις ε, πράσινες ε, τεχνολογίες 24 ε, επιχειρήσεις βρίσκονται στην Ασία, 22 στην Αμερική και μονάχα 4 ή 3 στην Ευρώπη. Επομένως θα πρέπει να το ξαναδούμε λίγο το θέμα αυτό γιατί η πράσινη οικονομία είναι ο νέος κλάδος της οικονομίας. Τώρα όσον αφορά αυτές τις διαρροές carbon leakage πολλά έγγραφα, πολύ μελάνη έχει χυθεί για το θέμα αυτό. Ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή, ε, αυτός ο ανοιχτός δρόμος ε, της ε, πράσινης οικονομίας αλλά ξέρουμε ότι και οι κίνδυνοι είναι μεγάλη. Όμως δυνητικά υπάρχουν τα εργαλεία και τα όπλα για να αμυνθούμε Επομένως ε, θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο τα κριτήρια ορισμού των ε, τομέων ε, κινδύνου και επίσης στη συζήτηση που θα κάνουμε μεταξύ μας θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε τι σημαίνει το πέρασμα στο 30%, τι σημαίνει να πάμε πέρα από το 20%. Ε, Υπάρχουν αυτές ε, οι, ε, αυτές οι πιστώσεις διοξιδίου του άνθρακα ε, και θα πρέπει να δούμε τι, σημαίνει, τι σημαίνουν ε, και επίσης να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε το πέρασμα στο 30% να είναι ένα πραγματικό και όχι ένα νοθευμένο πέρασμα. Ευχαριστώ πολύ. Η συνάδελφος Κόρχολα. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον άδελφο Ζόρδα Σίσελη για τις τόσο ισορροπημένες προτάσεις της. Ελπίζω σήμερα να μπορέσουμε να συζητήσουμε ε, τα αποτελέσματα της Κανκούν. Ήλπιζα τουλάχιστον αν δεν είναι δυνατό τι να κάνουμε. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στη Κανκούν δεν πετύχαμε αυτό που θέλαμε, δηλαδή ε, δεσμεύσεις για τη μείωση εκπομπών. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα όσα αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ε, καθώς επίσης και τη μετάβαση από το 20% στο 30% πλέον της αυτή όλη η συζήτηση για το 20-30% δεν εγγράφεται σε μια γενικότερη συζήτηση, ένα γενικότερο πλαίσιο. Και ποιο θα ήταν αυτό. Δεν έχει μελετηθεί, δεν έχει συντεθει καθόλου η αποτελεσματικότητα αυτών των μέσων και των μέτρων. Γιατί η ε, εμπορία ρήπων, ξέρετε, ότι μπορεί να λειτουργεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά έχουμε αποδείξεις πλέον ότι έγιναν πολλά σφάλματα μέχρι και απάτες στα πλαίσια αυτών των ανταλλαγών, των συναλλαγών της ε, αγοραπολισίας. Και αυτό έχει και επιπτώσεις στους ρήπους. Θελήσαμε λοιπόν να έχουμε μια περιοριστική πολιτική. Ωραία. Πολλοί όμως μεγάλοι ρηπαντές μας στέλνουν μηνύματα που λένε ότι δεν θέλουν να ποντάρουν εκεί, θέλουν να ποντάρουν στη γενοτομία, ε, στην ανανέωση, στην τεχνολογία, στην εξάλληψη του διοξιδίου του άνθρακα από την οικονομία. Είναι δύσκολο λοιπόν να συγκρίνουμε καταστάσεις και ε, ε, είναι και πολύ αργά για να συζητούμε τα 20-30%. Τώρα πλέον θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις μεγάλες αποφάσεις που μας περιμένουν. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να συγχαρώ πρώτα την εισηγήτρια για την ε, επιλογή του κειμένου. Θα πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί συμβιβασμός μεταξύ της Ήτρα και της ΕΜΠΗ και δεν θα είναι εύκολο υπάρχουν αυτοί οι οποίοι χαίρονται για τις διαπραγματεύσεις στο Κανκούν, άλλοι που έχουν εκ διαμέτρου ε, αντίθετο. Ε, αυτό είναι επίδειξη αισιοδοξία για μια συμφωνία που δεν υπάρχει. Τώρα το πέρασμα από το 20 30, χρόνια γίνεται λόγος αυτός. Εγώ θα ήθελα να γίνει μια αυστηρή αξιολόγηση του τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Τα μέτρα που πήραμε, τις συνέπειες που είχαν ε, και, στην, και όσον αφορά ε, μια οικονομία χωρίς διοξίδιο του άνθρακα, αλλά και όσον αφορά την ίδια την ανάπτυξη. Γιατί βρισκόμαστε σε μια πληρέστατη ασάφεια. Ας δούμε τι έχει γίνει, ας δούμε τι μέτρα έχουμε πάρει, ας δούμε τι εργαλεία έχουμε χρησιμοποιήσει, ας δούμε τη θετική πλευρά των εργαλείων αυτών, ας κάνουμε μια αξιολόγηση. Ας κάνουμε έναν απολογισμό ε, και ε, μετά να δούμε τι θα γίνει. Δεν θέλουμε ε, τον κανόνα της αμοιβαιότητας. Εμείς θέλουμε ό,τι κάνουμε εμείς απαρεγκλήτως να το ακολουθήσουν και οι άλλοι γιατί δεν έχει έννοια να έχουμε εμείς μία καθαρή οικονομία εάν στις άλλες υπήρους ε, που ξέρουμε ότι εκπέμπουν ε, ιδιαίτερα μεγάλα ποσοστά διοξιδίου του άνθρακος να μην ακολουθήσουν. Ε, και θα πρέπει όταν ε, θα ε, έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας, όταν θα έχουμε ήδη εφαρμόσει τα μέτρα, τότε οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουμε τον τρόπο και τους μηχανισμούς για να υποχρεώσουμε και τους υπολείπους να εφαρμόσουν το, τα ίδια συστήματα και ενδεχομένως ένα μηχανισμό αποκλεισμού στα σύνορα. I didn't understand. Yeah. Yeah. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη ε, συνάδελφο only to stress one point as για την καλή έκθεση και επειδή έχω ένα λεπτό μόνο ε, θέλω να πω το εξής. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να αναλύσουμε τις λύσεις για τους διάφορους κλάδους όπου υπάρχει κίνδυνος να σηκωθούν να φύγουν οι βιομηχανίες που παράγουν με πολύ διοξίδιο του άνθρακα. Εντάξει το 30% αλλά να τους προσφέρουμε και κάποιες λύξεις, να μην το διώξουμε αυτό τον κλάδο από την Ευρώπη. Υπάρχουν λύσεις, ε, λεγόμενες εγκάρσεις, προσεγγίσεις, ολιστικές, ό,τι θέλετε. Ε, σήμερα ας πούμε στο πρωτόκολλο του Κιώτο ε, τα δάση ή η πολιτική αεροπορία, ε, αερομεταφορές έχουν διαφορετική μεταχείριση. Δεν υπάρχουν στόχοι εθνικοί για μείωση, αλλά εγκάρση, οριζόντι. Θα μπορούσαμε λοιπόν, θα έπρεπε να μας απασχολήσει και αυτό για να δούμε αυτούς τους κλάδους που κινδυνεύουν να φύγουν από την Ευρώπη εάν παράγουν πολύ διοξίδιο του άνθρακα. Το είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Ε, υπάρχουν εθελοντικές συμφωνίες. Τα βέλη του ΕΛΚ εμείς τα μελετούμε και εγώ με την Πιλάρα και Αγιούσο και κάποιους άλλους. Καλό είναι να αφιερώσουμε κάποιο χρόνο στην εξέβριση λύσεων για αυτόν τον τομέα και να αναλύσουμε τις διάφορες πολιτικές. Είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία αυτά και για τη συζήτηση αυτή, αλλά και για άλλες, για τις μελλοντικές. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος λάγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα επιπλέον σημείο, αν μου επιτρέπετε, κυρία Συγήτρια, θέλω να βάλω εδώ και μια χρονική διάσταση. Αν κοιτάξουμε ρεαλιστικά, είμαστε τώρα στο 2011. και πριν ε, είναι στο στάδιο της εφαρμογής τα μέτρα θα περάσουν δύο-τρία χρόνια τουλάχιστον. Οπότε δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο να σκεφτούμε και περαιτέρω μείωση. Και το λέει και έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη σελίδα 1. Καλό θα ήταν ήδη από τώρα να προσανατολισόμαστε για το 2050 παρακαλώ για να έχουμε πιο μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Γιατί σήμερα τι γίνεται. Πολλοί κλάδοι της οικονομίας, της βιομηχανίας δεν ξέρουν τι θα ε, κάνουν, ποια θα είναι η περίοδος για ε, τις εκπομπές και το εμπόριο ρήπων γιατί δεν έχουμε ακόμα τη συγκριτική αξιολόγηση, το benchmark και δεν μπορούμε να ερχόμαστε μετά από δύο-τρία χρόνια να τα ε, ανατρέπουμε αυτά. έτσι, να σκεφτούμε το πλαίσιο ευρύτερα και πιο μακροπρόθεσμα. Ο συνάδελφος Μεσάρος. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέκαθεν αγωνιζόταν κατά της κλιματικής αλλαγής και προσπαθούσε να την καταπολεμήσει. Νομίζω ότι ε, ο στόχος του να περάσουμε από το 20% στο 30% είναι κάτι το οποίο έχει ξεπεραστεί από τις εξελίξεις. Έχουμε πλέον την οικονομική κρίση που πλήττει και τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Και παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εγκαταλείπει, δεν απεμπολεί αυτή την προσπάθεια κατά πολέμης κλιματικής αλλαγής. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το στόχο του 20% πρώτα τι σημαίνει, αν μπορούμε να τον πιάσουμε και μετά να εξετάζουμε την ε, ιστορία του 30%. Και αυτό θα ε, είναι πολύ χρήσιμο και για τη βιομηχανία μας και θα μπορέσει να επενδύσει αλλού σε θέσεις απασχόλησης για παράδειγμα. Και να είναι αυτή μια ευρωπαϊκή στρατηγική. Γνωρίζουμε ότι ο κόστος στρατηγικής 2020 έχει μεν μειωθεί, αλλά πρέπει να συζητήσουμε από τώρα τις επιπτώσεις όλων αυτών των αλλαγών και το να γίνει 20-30%. Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να γίνει αυτό από τώρα. Ε, πρέπει να τις δημιουργήσουμε. Συνδεόμαστε με διεθνείς εταίρους, συνεργαζόμαστε. Θα πρέπει να βρούμε ε, κίνητρα. Κάθε χώρα να κάνει και άλλες προσπάθειες. Γι' αυτό είναι σημαντικότατη η διεθνή συνεργασία. Και απαραίτητη. E, panie Przewodniczący, ja myślę i bardzo popieram to, co powiedziała Pani. Mm, e, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ πάρα πολύ ε, και υποστηρίζω αυτά που είπε η κυρία Τζόρνταν. Δηλαδή, θα πρέπει να κάνουμε ακρόαση, να καλέσουμε εμπειρογνώμονες που γνωρίζουν ε, πάρα πολύ καλά συγκεκριμένες περιφέρειες. Γιατί έχουμε αυτή την τάση συχνά να ε, ψάχνουμε λύσεις και να υιοθετούμε λύσεις κατά ε, για όλους. Μα δεν γίνεται αυτό. Είναι διαφορετικές οι εθνικές οικονομίες, είναι διαφορετικά κράτη. Δεν μπορούμε να αλλάζουμε έτσι τα όρια αβίαστα. Ακόμα και ε, για ένα μικρό ποσοστό, αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιες χώρες. Υπάρχουν χώρες που βασίζονται πάρα πολύ στον άνθρακα. Ε, για τις ενεργειακές τους ανάγκες. Δεν μπορούν να εξισώνονται όλες οι χώρες, δεν είναι στην ίδια μοίρα. Και πώς θα περάσουμε από το 20 στο 30, μήπως να λέγαμε 25% για χώρες που εξαρτώνται πάρα πολύ από τον άνθρακα. Και αυτό το θέμα στην Πολωνία είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η απειλή να σηκωθούν να φύγουν οι βιομηχανίες, δηλαδή αυτό το carbon leakage. Ενώ έχουμε ξένες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, το, το άνθρακα μας απειλούν ότι θα σηκωθούν να πάνε στην Ουκρανία. Γιατί είναι πάρα πολύ υψηλό το κόστος των στόχων που θέτουμε. Και τι θα λυθεί το πρόβλημα αν πάνε να φτιάξουν εργοστάσιο στην Ουκρανία. Οι ρήποι δεν γνωρίζουν σύνορα, στην ίδια Ήπειρο βρισκόμαστε. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με χώρες ε, ε, παραμεθόρια, δηλαδή με τις οποίες συνορεύουμε και μπορούμε να τις επηρεάσουμε πολιτικά και οικονομικά. Και δεν είναι κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Η συγκητρία. Θες να πεις τίποτα? Σύντομα σε παρακαλώ. Ναι, ναι. <clears throat> Θα ήθελα να σχολιάσω, αλλά δεν μπορώ να σχολιάσω βεβαίως κάθε παρέμβαση. Πάντως είμαι ευτυχής ε, γιατί ε, θα δούμε πλέον σε αυτήν την ε, θητεία πώς θα εφαρμόσουμε κάποιες νέες αρχές και επίσης πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα μέχρι το 2020 ενδεχομένω και ε, συμφωνώ με τους συναδέλφους που ανέφεραν το 2050 ως χρονικό ορίζοντα και όχι το 2020. Είναι γεγονός ότι μας λείπουν κάποια ε, στοιχεία και επομένως χρειαζόμαστε ε, πληροφόρηση. Αυτό θα γίνει μέσω ακρόασης είτε εάν συνδυαστούμε με την Επιτροπή Περιβάλλοντος είτε και εάν χρειαστεί να κάνουμε δική μας ακρόαση. Επίσης να δούμε τον ρόλο των περιφερειών ε, και η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι βλέπει μεγαλύτερες δυνατότητες ε, εάν επικεντρωθούμε και στις πιο φτωχές χώρες. Πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτό για μας. Όσον αφορά την ψηφοφορία ε, για την, στην Ολομέλεια θα πρέπει να συμφωνήσουμε και με τον Επιτροπή και με την Επιτροπή, με τον εισηγητή δηλαδή της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος φοβούμε ότι δύσκολα θα μπορέσουμε να προλάβουμε ε, πριν από τον Μάιο. Το Μάιο θα πάρει την απόφαση στο Συμβούλιο. Δύσκολο να προλάβουμε να ψηφίσουμε πριν τον Μάιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ αρκετά γρήγορα να ξεκαθαριστεί αυτό το θέμα τη ακρόαση. Αν μπορούμε να κάνουμε κοινή ακρόαση και αν όχι εμεί το συντομότερο να φροντίσουμε να το προωθήσουμε όπω ζήτησαν πολλοί συνάδελφοι. Ωραία. Πάει και αυτό το θέμα στη μέρησια διάταξη. Θα παρακαλούσα τώρα το 10 να το αναβάλουμε γιατί έχει έρθει ο προσκεκλημένος. Περιμένει εδώ και ένα τέταρτο και ε, δύο είναι τα τεινά τώρα. Είτε θα συζητήσουμε το θέμα του κυρίου Αντάμοβιτς και μετά θα ασχοληθούμε με την Κανκούν είτε θα αναβάλουμε την Κανκούν για την επόμενη συνεδρίαση και τα δύο γίνονται αλλά να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Δεν έχω πρόβλημα, θα εξαρτηθεί και από τους ε, ενδιαφερομένους να το αναβάλουμε για την άλλη φορά. Λένα Εκ, next time, καλώς. Όλοι θέλετε Γι' αυτό έχουμε τρία τέταρτα τώρα να ασχοληθούμε με το άλλο θέμα, με την ησυχία μας. Ζητώ συγγνώμη. Δεν ξέρω, μετά τις διακοπές έχουμε χαλαρώσει ή φορτώσαμε πολύ την ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω λοιπόν τον κύριο Αντάμοβιτς. Καλωσορίσατε. Είναι ο Ευρωπαίος Συντονιστής για τη Συνδέση με το Δίκτυο Υλικής Ενέργειας Ανοιχτής Θαλάσσης στη Βόρεια Ευρώπη έχει μια έκθεση να μας παρουσιάσει και έχουμε και ευκαιρία εμείς να του κάνουμε ερωτήσεις. Καλώς ορίσατε πρώτα απ' όλα. Κυρία ε, Αντάμοβιτ, σας εύχομαι καλή χρονιά, ε, καλή δύναμη. Έχετε το λόγο μόνο εσείς και κανένα άλλος και παρακαλώ όλους τους συναδέλφους να κάνουν ησυχία και να ακούσουμε προσοχή. Να είστε κι εσείς σαφής, περιεκτικός, συνεκτικό, εύστοχος, όπως ξέρετε πάντα να το κάνετε και μετά να εκμεταλλευτούμε το χρόνο για τη συζήτηση. Ναι, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας μιλήσω ως συντονιστής για τις συνθέσεις με το δίκτυο ολικής ενέργειας ανοιχτής θαλάσσης στη Βόρεια Θάλασσα και στη Βαλτική. Σας έχω στείλει ε, την ομιλία μου, την έκθεσή μου, δεν θα τη διαβάσω γι' αυτό. Στην Ευρώπη των 27, με τα 400 περίπου 50 εκατομμύρια κατοίκους, ε, ε, ξέρω ποια είναι η δική μου δουλειά, η δική μου αποστολή. Προβληματίστηκα, είναι δυνατόν εγώ να λειτουργήσω σε μια τόσο μεγάλη κλίμακα. Πάντω πήγαν πολύ καλά τα πράγματα. Ε, έχω πολύ μεγάλη υποστήριξη από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργεια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω ένα συνεργάτη, έναν υπάλληλο ε, δικό του και προχωρήσαμε πολύ και για εσάς είναι σημαντικό αυτό γιατί ε, συζητήσατε για χρηματοδότηση. Ο Ευρωπαίος Συντονιστής δεν έχει ιδίους πόρους, πράγμα που δυσκολεύει πάρα πολύ τη δουλειά μας επί τόπου γιατί ε, αν χρειαζόμαστε να παραγγείλουμε μία αντικειμενική μελέτη από την άλλη όταν κάποιος ε, δεν χρηματοδοτείται από ένα δημόσιο κορβανά είναι πιο ελεύθερο στη σκέψη του, στη δράση του γιατί δεν περιορίζεται από τη χρήση του δημοσίου χρήματος ε, μηνιαία βέβαια έχω ε, κάποιο μισθό από την Ευρωπαϊκή Ένωση αρκετά πενιχρό σε σχέση με τα όσα περιμένουν από μένα και μου έχουν αναθέσει. Ε, πρέπει να το πω και αυτό. Η Ευρώπη είναι πάντα πάρα πολύ φιλόδοξη, αλλά όταν πρόκειται για ποιότητα είναι λίγο περιορισμένη και στα οικονομικά της. Αυτά. Ποιο είναι τώρα το έργο του συντονίστη. Ε, συνέστησα μια ομάδα εργασίας η οποία στο μεταξύ ασχολείται με τις χώρες της Βόρειας Θάλασσας και της ε, Βαλτικής και είναι εγκατεστημένη εκεί. Είναι πάρα πολύ άτυπη. Εκπροσωπείται η πολιτική, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε εκεί διάλογο. Η ιδιωτική οικονομία, έτσι ώστε να έχουμε τι διάφορε διαφορετικέ απόψεις, μια εικόνα πλήρη για όλα τα θέματα και διαβιβάζονται αρμοδίω και αυτά. Συνεδριάζει η ομάδα εργασία αυτή τουλάχιστον κάθε τρίμηνο στι ε, Βρυξέλλε και αλλού και ε, είναι και βασικός χώρος της εργασίας μου. Κατά τα άλλα έχω επαφές με κυβερνήσεις, με την κοινωνία των πολιτών κτλ το εργαλείο, το μέσο που έχω στη διάθεσή μου είναι η ετήσια έκθεση μου που πρέπει να υποβάλω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από τα τέλη του έτους έχετε εσείς στα χέρια σας την τρίτη αυτή η έκθεση και θα σας παρουσιάσω λίγο τα αποτελέσματά της. Πρώτον, γενικά. Όταν γίνεται λόγος για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρώπη, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι χωρίς διεύρυνση και τροποποίηση ε, των ε, σημερινών υποδομών και δικτύων, αυτό δεν γίνεται. Αυτό αφορά τους φιλόδοξους στόχου της Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά για να γίνουν πραγματικότητα αυτοί θα πρέπει ουσιαστικά να ασχοληθούμε με την υποδομή ενέργειας. Εδώ κυρίως μιλώ για την ηλεκτρική ενέργεια και να ασχοληθούμε περισσότερο. Στις συζητήσεις που είχα στις διάφορες χώρες και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και παντού γίνεται λόγος για τις εξουσίες και αρμοδιότητες της Ευρώπης ε, πολύ περιορισμένα όμως για τη διεύρυνση και την επέκταση των δικτύων. Είναι το άρθρο 194 ε, της Συνθήκης Λισαβόνας που ορίζονται καταρχήν οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόλις αναφέρει κανείς αυτό το άρθρο εκπλήσονται οι πάντε γιατί δεν το γνωρίζει κανείς αυτό. Και ιδιαίτερα το θέμα της μεταφοράς, της ενέργειας των δικτύων μεταφορών είναι όλο και περισσότερο πλέον ευρωπαϊκό θέμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό το πρώτο αυτό για μένα. Θα πρέπει πολύ περισσότερο να δεσμευτούμε προς την κατεύθυνση αυτή και να τονίζουμε ότι έχει η Ευρώπη αρμοδιότητες γιατί έτσι δικαιολογείται και η ανάγκη και πολιτικά και οικονομικά να ε, αναπτυχθούν δίκτυα στην Ευρώπη. Αυτό ισχύει και για την ανοιχτή θάλασσα αλλά και για τις ε, εγκαταστάσεις στην ξηρά. Έχουμε στόχους στην Ευρώπη για το κλίμα, το στόχο του 20% ας πούμε. Τι σημαίνει αυτό, το 2020 να έχουμε 20% μερίδιο ε, των ανανεωσίμων στον ηλεκτρισμό αυτό είναι 35%. Καλή είναι η συζήτηση τώρα για το 30%. Αν το 20% όμως γίνει 30% χωρίς ε, χρονικό ορίζοντα και ε, στον ηλεκτρισμό είναι πάνω από το 50% αυτή η αναλογία, το μερίδιο. Τι σημαίνει αυτό. Τίποτα παραπάνω παρά βιομηχανική επανάσταση. Είναι τίποτα διαφορετικό μάλλον. Και ε, χρειάζεται τελείως διαφορετική πολιτική για να φτάνει αυτό το παραγόμενο προϊόν στον καταναλωτή. Αν δούμε τι δυναμικό έχει η Βόρεια Θάλασσα και η Βαλτική, για το 2020 είναι 40 γιγαβάτ και το 30 150 γιγαβάτ το δυναμικό που θα μπορούσαμε να εξαντλούμε. Αυτά είναι τεράστια μεγέθη. Ε, με μεγάλες ευκαιρίες, αλλά για να επιτύχουν θα πρέπει όχι μόνο να κάνουμε ολικά πάρκα, αλλά να φέρνουμε και το παραγόμενο προϊόν, το ρεύμα στον καταναλωτή 24 ώρες το 24ωρο. Συγκεκριμένα τώρα σημεία της έκθεσής μου. Είναι καλό και ευχάριστο να μιλάμε για επιτυχίες, αλλά θα ήθελα να αρχίσω από ένα θέμα που είναι ευρωπαϊκή πανολεθρία. Και είναι το έργο Κρίγας Φλακ στην ε, Βαλτική όπου συμμετέχουν τρεις χώρες, συμμετείχαν Γερμανία, Δανία, ε, Σουηδία για να αντιληφθεί όσο γίνεται περισσότερο δυναμικό από τη Βαλτική και δυστυχώς κατά τη διάρκεια ε, της Σουηδικής Προεδρίας η Σουηδία αποχώρησε από το έργο για τη συζήτηση αυτή των αιωλικών πάρκων στη θάλασσα είναι σημαντικό αυτό. Γιατί πραγματικά αυτή η τριεθνή συμμετοχή θα εξασφάλισε απαντήσεις σε πολλά σημαντικά ζητήματα ω προς την ανάπτυξη της αγοράς, τεχνικά ζητήματα και πολλά άλλα. Έτσι, ένα τριεθνές πρόγραμμα ε, ευρωπαϊκό και δυστυχώς ε, στο, η φάση ακόμα του προγραμματισμού αποχώρησε μία από τις τρεις χώρες. Κρίμα. Και πραγματικά το λέω... Ε, ε, ότι είναι καταστροφή η πανολεθρία στα μέσα της Βαλτικής. Αν καταλάβουμε ε, ότι χρειάζονται διασυνδέσεις ε, οι υποδομές στην Ευρώπη, αν θέλουμε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο. Μας λείπει αυτή η διασύνδεση τώρα και θα ήταν χρήσιμο και απαραίτητο όχι μόνο για την Νορβηγία αλλά και για τη Σουηδία να έρθει πιο κοντά στην κεντρική Ευρώπη. Κρίμα, κρίμα που και στη δημόσια συζήτηση και στην πολιτική συζήτηση δεν εμφανίζονται αυτά τα προβλήματα. Δεν μας απασχολούν. Δεν θα πρέπει να αναρωτηθούμε προς τα πού πηγαίνουμε στην Ευρώπη. Εύκολο είναι να ορίζει στόχους, η υλοποίηση είναι δύσκολη. Και αν φτάσουμε σε ένα τέτοιο έργο δεν είναι καλό επισκεπτήριο, δεν είναι ε, διαφήμιση για την Ευρώπη αυτό. Σε αυτά τα λόγια δεν θέλατε σταράτα από τον Ευρωπαίο Συντονιστή, ειδού. Επιτυχίες τώρα, κυρίες και κύριοι η 7η Δεκεμβρίου του 2010. Γιατί οι 10 χώρες της ε, Βόρειας Θάλασσας, συμπεριλαμβανομένης και της Νορβηγίας, υπέγραψαν ένα μνημόνιο συνεννόησης ε, με τρία θέματα συνεργασίας. Το ένα είναι η εξήγηση τεχνικών ζητημάτων του δικτύου της Βόρειας Θάλασσας, το δεύτερο προβληματισμοί για την αγορά, πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί μια μελλοντική αγορά και επίσης ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ηλεκτρικό ρεύμα δηλαδή καλύτερα στην αγορά αυτή και το τρίτο ε, θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού και έγκρισης. Σε ένα μνημόνιο λοιπόν ε, συνεννόησης ε, καταγράφηκαν αυτά για μια διετία και το 2012 θα καταλήξουν οι εργασίες για αυτές τις 10 χώρες και θα έχουμε μια εκτίμηση για το ποιες είναι οι προϋποθέσεις εκείνες που πρέπει να δημιουργηθούν ε, στο δίκτυο οικονομικά και ε, γενικότερα για να γίνει πραγματικότητα ο ευρωπαϊκός στόχος. είναι πραγματικά υπόδειγμα και επικεντρώθηκα και εγώ πάρα πολύ σε αυτό και είναι μεγάλη επιτυχία που οι 10 αυτές χώρες συμφώνησαν, συνεννοήθηκαν. Γιατί λέω ότι είναι μεγάλη επιτυχία, διότι και οι εταιρείε ε, που έχουν αναλάβει τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας συμμετέχουν και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές οι εκάστοτε. Η ρυθμιστική αρχή ενέργεια είναι μια ευρωπαϊκή εφεύρεση, εντάξει κανένα πρόβλημα. Ε, κυριαρχεί ε, σε αυτό το θέμα της ε, επέκτασης, εξάπλωση και ανάπτυξη του δικτύου, αλλά χρειάζεται πολιτική καθοδήγηση. Ευρωπαϊκή, πολύ περισσότεροι αυτοί οι εθνικοί ρυθμιστικοί οργανισμοί. Γι' αυτό Λοιπόν, στη Βόρεια Θάλασσα ήταν ε, το μεγαλύτερο επίτευγμα των τελευταίων ετών αυτό. Δεύτερη παρατήρηση για το ίδιο θέμα, για μια που αναφέρθηκα στις ρυθμιστικές αρχές. Νομίζω ότι στην Ευρώπη θα πρέπει να γίνει μια πολύ πιο εντατική συζήτηση ε, ουσιαστική με τις ρυθμιστικές αρχές. Πολλές φορές ε, είναι υπερβολικά προσιλωμένες και προσδεμένες σε εθνικές ε, νομοθεσίες και η αδειοδότηση των νέων δικτύων δεν λαμβάνει αρκετά υπόψη ε, τις επενδύσεις στο κεφάλαιο, γιατί κάθε ρυθμιστική απόφαση καθορίζει και προσδιορίζει τη δυνατότητα κεφαλαιακής παρέμβασης ε, των εταιριών οι οποίες εταιρείε όμως θα πρέπει να αντλήσουν κεφάλαια από τις αγορές και η ρυθμιστική αρχή τους υπαγορεύει τι κέρδο θα έχουν από αυτή την επένδυση και τους το επιβάλλει. Ε, αυτό ισχύει και για δημόσιες ε, εταιρείε, ε, αλλά και για ιδιωτικές που διαχειρίζονται το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας. Τα χρήματα τα παίρνουν από τις αγορές. Και όταν φτιάχνει κάποιος ε, μία σύνδεση με τρει-τέσσερι χώρε α πούμε, στη Βόρεια Θάλασσα, όπου παρεμβαίνουν τρει-τέσσερι ρυθμιστικέ αρχές, αυτό έχει αρνητικέ επιπτώσεις στα δάνεια, στην επένδυση, στο, επιτόκιο που θα δώσουν οι αγορές ε, στην επιχείρηση. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ε, οικονομική ε, πρόκληση. Ε, τι γίνεται με το πλαίσιο το ρυθμιστικό των χρηματαγορών και πώς θα καταφέρουμε ακριβώς αυτές οι αρχές να ε, έχουν μια πολύ πιο ευρωπαϊκή νοοτροπία και όχι εθνική στις αποφάσεις τους. Το αναφέρω και στην έκθεσή μου. Θα μπορούσα να φανταστώ εδώ να έχουμε πιο ευρωπαϊκή λύση και να συσταθεί μια ομάδα τετραμελής, πενταμελής στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να μελετά αυτό το θέμα για τις ενεργειακές επενδύσεις πώς επιδρούν στις χρηματαγορές ε, οι ρυθμιστικές αρχές με τις αποφάσεις τους χωρίς να συμμετέχουν οι ρυθμιστικές αρχές αλλά να ε, απαντούν αν δέχονται ή αν δεν δέχονται τις υποδείξεις Εθνικής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό θα έφερνε μεγαλύτερη διαφάνεια χωρίς πολύ μεγάλη διαρθρωτική αλλαγή, ένα πακέτο για την εσωτερική ενιαία αγορά κτλ. όπου ορίζονται οι αρμοδιότητες των ρυθμιστών. Χωρίς να δημιουργηθεί νέα γραφειοκρατία, μια χρήσιμη συμπλήρωση θα ήταν κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εκεί χρειάζεται να ενταθούν οι προσπάθειες και να είναι πιο διαφανής οι αποφάσεις που παίρνουν οι ρυθμιστικές αρχές απέναντι στην κοινή γνώμη, την πολιτική, γιατί είναι πάρα πολύ φιδωλή ε, στην ενημέρωση. Το επόμενο, όταν μιλεί κανείς και με τους ενδιαφερόμενους, το offshore δεν έχει νόημα αν δεν υπάρχει και η σωστή διασύνδεση. Είναι τα προβλήματα σχεδιασμού που έχουμε στην Ευρώπη. έχουμε μια ευρωπαϊκή σύγκρουση εδώ. Θα την εξηγήσω. Από τη μια μεριά έχουμε μια ιδιαίτερα δεσμευμένη πολιτική ενέργειας που ρίχνει μεγάλο βάρος στις εναλλακτικέ ενέργειες. Βεβαίως δεν υπάρχει άλλη λύση, αυτό είναι γεγονός, συμφωνούμε. Όμως αντιμετωπίζουμε μεγάλα προβλήματα έγκρισης, αδειοδότησης όταν έχουμε προβλήματα υποδομών, έργα δηλαδή υποδομών. Από την άλλη μεριά έχουμε και μια πολιτική προστασία της φύσης, Natura κλπ. Και εδώ κάπου έρχονται και συγκρούονται δύο ευρωπαϊκές αηφόρες στρατηγικές. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν και οι σωστές διασυνδέσεις, η αγωγή. ...42 χιλιάδες χιλιόμετρα γραμμές υψηλής τάσος. Εγώ ο ίδιος δεν μπορώ να κρίνω τον αριθμό αυτό, ίσως είναι και υπερβολικά υψηλό. Πρόκειται για τεράστιο έργο που θα επηρεάσει και τους στόχους προστασίας του κλίματος κτλ. Λοιπόν, ε, σας εξήγησα την αντίφαση. Πώς αντιμετωπίζουμε την αντίφαση. Εγώ ζήτησα και έγινε μια πραγματογνωμοσύνη που τη βάζω ε, παράρτημα στην έκθεσή μου. Η πραγματογνωμοσύνη καταλήγει ότι δεν υπάρχει κανένας χώρος να παραιτηθεί η Ευρώπη από τις διάφορες οδηγίες προστασίας της φύσης, ε, της τη χλωρίδα κτλ. Αλλά ίσως χρειάζεται διαφορετική ε, θέσπιση προτεραιοτήτων. Και η λύση που προτείνω εγώ έχει ως εξή να συμπληρωθούν οι οδηγίες προστασίας των κτηνών και FFA με την έννοια δηλαδή ότι όταν ένα έργο κατασκευής γραμμών υψηλών τάσεων συνδυάζεται με την στρατηγική της, ε, των ανανεώσιμων πηγών και ούτω καθεξής θα πρέπει να έχει η γραμμή υψηλής τάσεως προτεραιότητα απέναντι σε ορισμένες από τις ανάγκες προστασίας της ε, οδηγίας προστασίας χλωρίδας και πανίδας κλπ. Από την επαγγελματική μου εμπειρία δεν έχει νόημα να παράγουμε πράγματα τα οποία διαρκώς πρέπει να τροποποιούνται. Έκανα μία πρόταση, την οποία συνοδεύω και με μία πραγματογνωμοσύνη, με ευρωπαϊκή θεμελίωση και τουλάχιστον θέλω να συζητηθεί. Δεν έχει νόημα δηλαδή να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας αν δείτε την κατάσταση στα σύνορα μεταξύ Γερμανίας και Βελγίου, τι θα γίνει στο, στα επόμενα 5-6 χρόνια εάν βγει η ΕΣΑ και πει ότι χρειαζόμαστε ένα νέο, ε, μια νέα διασύνδεση μεταξύ των δικτύων Γερμανίας και Βελγίου ενώ ταυτόχρονα ολόκληρη αυτή η περιοχή βρίσκεται υπό ε, καθεστώς προστασίας. Δεν περνάει από εκεί με τις παρούσες συνθήκες, με τις παρούσες ρυθμίσεις γραμμή υψηλής τάσος τι θα κάνουμε μετά με άλλο. Το Τέζα Τεκ, με το οποίο ίσως θα μπορούσαμε να επιτύχουμε τα 20% με το 2050. Πώς, τι θα κάνουμε στα Πυρηναία, όπου ήδη σήμερα η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη σε ό,τι αφορά τη δημιουργία γραμμών υψηλή τάσο. Εδώ βρίσκονται οι συγκρούσει, εδώ βρίσκονται οι αντιφάσει. Πρέπει να συζητηθούν πολύ εντατικότερα δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Πρέπει στην Ευρώπη να έχουμε την διάθεση να συζητήσουμε και μάλιστα πολύ επιθετικότερο τρόπο τις ε, αντιφάσεις αυτές. Στην πραγματογνωμοσύνη αυτή περιλαμβάνεται μία φράση που λέει ότι η Ευρώπη δεν επιτρέπεται να αφήσει τις χώρες ε, στη μοίρα τους, τις χώρες μέλη στη μοίρα τους σε αυτό το θέμα. Βρίσκω λοιπόν αξιοσημείωτη τη φράση αυτή. Τώρα για να μην είναι θεωρητική η προσέγγιση Έχω περιλάβει 7 έργα τα οποία έχουν ευρωπαϊκή διάσταση και από τα ε, προγράμματα δηλαδή των ε, ευρωπαϊκών δικτύων, ευρωπαϊκών δικτύων, όπως είπα, χρειαζόμαστε από τον σχεδιασμό μέχρι την κατασκευή μιας γραμμής υψηλής τάσης χρειαζόμαστε από 10 έως 15 χρόνια. Έχουμε όμως το στόχο μέχρι το 2020 να έχουμε 25% ε, μετακίνηση της ενέργειας προς την ηλεκτρική ενέργεια. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Το επόμενο θέμα πρέπει να ασχοληθούμε πολύ περισσότερο με τα τεχνικά θέματα. Εναλλασσόμενο ρεύμα, μη εναλλασσόμενο ρεύμα. Τι γίνεται όμως διεξάγεται διάλογος, καρποφόρος διάλογος και με τις επιχειρήσεις και κύριε Πρόεδρε, νομίζω να εξετάσετε εάν ίσω από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια των πιλωτικών προγραμμάτων. Δεν θα πω περισσότερο σε τεχνικά θέματα γιατί δεν έχουμε τον απαραίτητο χρόνο. Όταν όμως μιλούμε για την αναγκαιότητα ευρωπαϊκών αγωγών θα μιλήσω και για την αναγκαιότητα ευρωπαϊκών πιλωτικών προγραμμάτων για να τεθούν επιτάπητος τεχνολογικά προβλήματα να συζητηθούν, να προκύψουν λύσεις που είναι σημαντικά και για, την, για να αποτελέσουν τη βάση για τις ρυθμιστικές αποφάσεις. Εγώ περιλαμβάνω πολλές προτάσεις για το πώς θα πρέπει να διαμορφωθούν αυτά τα πράγματα ή πώς μπορούν να διαμορφωθούν. Το επόμενο που έχει σχέση με σχεδιασμό και αδειοδότηση είναι η εμπειρία που έχω από το έργο Ζάλτσπουργκ όπου με συμμετοχή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ορίστηκα ως Ευρωπαίος Συντονιστής και πέρασα 6 μήνες τον προηγούμενο 1,5 χρόνο στην Αυστρία και μπόρεσα να προωθήσω ένα έργο το οποίο είχε καταλήξει σε αδιέξοδο τα τελευταία 10 χρόνια. Ένα πρόβλημα που είχε προκύψει ήταν το θέμα θα είναι ε, υπόγειο καλώδιο ή ε, ένα αέριο. Πολλά τεχνολογικά προβλήματα μπορούσαν να συζητηθούν. Η τεχνολογία της, ε, του ελεύθερου αγωγού δεν είναι ίδια με το καλώδιο. Δεν έχει κανένα νόημα όμως να καταδικάσουμε τη μία τεχνολογία και να ε, θεοποιήσουμε την άλλη. Πρέπει να συζητήσουμε και θέματα αριθμιστικά, εάν δηλαδή εν μέρη χρησιμοποιήσουμε καλώδιο, μπορεί ένα μέρος το κόστος να μετακυλιστεί στους τελικούς καταναλωτές. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, πρότεινα στο θέμα αυτό το οποίο οδήγησε και σε πολύ αντιφατικές συζητήσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθίσει να συζητήσει με τους Ευρωπαίους κατασκευαστές καλωδίων. Πήγε πολύ καλά αυτή η διαδικασία, τα γράφω στην έκθεσή μου, προέκυψε έγγραφο συνένεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαίων κατασκευαστών καλωδίων, ώστε τουλάχιστον να έχουμε κάτι στα χέρια μας, για να μπορέσει να γίνει και μια συζήτηση αξιολόγησης και να μην υπάρχει αιμονή σε ορισμένα επιχειρήματα εκατέρωθεν διότι είναι, είναι πράγματι σκόπιμο να συζητηθεί το θέμα. Μιλώντας τέλος για εναλλακτικέ ενέργειες και πάλι επανέρχομαι στο θέμα της Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής και με το συνδυασμένο τους δυναμικό καταλήγω στο ότι στην Ευρώπη πρέπει να συζητήσουμε πολύ περισσότερο τα περιφερειακά δυναμικά, τα οποία δεν συμμετέχουν στα εθνικά δίκτυα. Η Βόρεια Θάλασσα είναι πολύ εθνική περιοχή, μέχρι και τη Σκωτία. Είναι σαφές λοιπόν ότι αν εξεταστεί έτσι, στην ουσία σημαίνει ανάγκη μιας άλλης ευρωπαϊκής συζήτησης. Το καθιστώ σαφές αυτό στην έκθεσή μου με ορισμένα παραδείγματα, γιατί είναι σαφές ότι βγαίνοντας στις θάλασσες βλέπουμε ότι οι μεν κάνουν το ένα πράγμα, οι άλλοι κάνουν άλλο πράγμα. Οι εναλλακτικέ ενέργειες έχουν και ένα μέγα οικονομικό δυναμικό. Τα συζητήσατε σήμερα αυτά. Καταλήγει κανείς τότε στο συμπέρασμα ότι τα θέματα αυτά στην Ευρώπη πρέπει να συζητηθούν διαφορετικά και από την οικονομική ε, σκοπιά και από την σκοπιά διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος. Σε αυτό που κάνουμε τώρα από πλευρά συντονισμού παρακολουθούμε την διαδικασία αυτή στην οποία αναμειγνύονται 10 χώρες που βρέχονται από την Βόρεια Θάλασσα. Έχουμε και ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα για το τι θέλουμε να κάνουμε φέτος. Στην διάρκεια του φετινού χρόνου θα κριθεί κιόλας εάν θα ανανεωθεί η εντολή μου η οποία λύγει ναι, εντάξει, έτσι είναι τα πράγματα, normal είναι αυτό. Εγώ έχω... Ε, βλέπω τον κύριο Τούρμες που γελά. Ε, μου άρεσε η εργασία που έκανα. Συνέβαλα και σε μια μεγαλύτερη διαφάνεια σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ε, σας ευχαριστώ λοιπόν που με παρακολουθήσατε. Ε, σας συνιστώ να διαβάσετε την πραγματογνωμοσύνη. Ευχαρίστω να έλθω στι πολιτικέ σα ομάδε να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Περιλαμβάνονται πολλές λεπτομέρειες και για τα θέματα ε, διαδικασίας ε, σχεδιασμού και αδειοδοτήσεω που έχει πολύ θα έλεγα είναι θέμα ακαθόδες, έχει πολύ εκρηκτικό δυναμικό δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς ιδιαίτερα τις ε, οδηγίες ε, προστασίας περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ κύριε Αντάμωβιτς πρώτα για την εργασία σας. Αυτό είναι αυτονόητο. Δεύτερο, και για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάσατε το θέμα σας. Το βρήκα ιδιαίτερα ενδιαφέρον που θέσατε τα προβλήματα και που προτείνετε και λύσεις. Και δεν αρκεστήκατε μονάχα στο να μας παρουσιάσετε έναν όμορφο κόσμο αγγελικά πλασμένο. Το αν θα ε, συμφωνήσουμε ή όχι μαζί σας αυτό είναι ανοιχτό. Τουλάχιστον όμως έχουν τεθεί τα προβλήματα. Και ότι υπάρχουν ενδεχόμενες λύσεις. Αυτό θα μας βοηθήσει πολύ. Σας ευχαριστώ λοιπόν ιδιαίτερα γι' αυτό και είμαι βέβαιος, απόλυτα βέβαιος, ότι κάποιες πολιτικές ομάδες θα θελήσουν να επανέλθουν στην, ε, να δεχθούν την πρόσκλησή σας δηλαδή για να συζητήσουν κι άλλο μαζί σας. Τώρα το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Τούρμες. Μάλιστα, ήταν πολύ ζωηρή η ε, παρουσίασή σας. Μου αρέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι μιλούν καθαρά. Είστε άλλωστε και κάποιος ο οποίος εργάζεται στον τομέα της ενέργειας από πολλά χρόνια. Δεν έχω διαβάσει δυστυχώς την έκθεσή σας με όλες τις λεπτομέρειες. Θα θέσω ωστόσο ορισμένα ερωτήματα, θα κάνω και κάποια σχόλια. Πρώτα σας ευχαριστώ που είπατε καθαρά ότι η ανανεώσιμη ενέργεια είναι η εναλλακτική επιλογή. Για το 30% μέχρι το 2020 δεν σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάμε στο 35% εναλλακτικές ενέργειες πιο πολύ για να γίνει η εξοικονόμηση αυτή πρέπει να μας απασχολήσει η αποδοτικότητα της φυστάμενης ενέργειας. Μιλήσατε και για τα μεγαβάτ της ε, Βόρειας Θάλασσας, Βόρεια Θάλασσα, Βαλτική Θάλασσα. Εκεί μπορούμε να κερδίσουμε στη συζήτηση που κάνουμε και για ανεξαρτησία ε, ενέργειας, γιατί εκεί έχουμε περισσότερη ενέργεια από ό,τι έχει ολόκληρη Ρωσία. Για το έργο Kriegers Φλακ» Σας ευχαριστώ που τα είπατε καθαρά. Για μένα είναι πολύ κακό παράδειγμα αυτό που έδωσαν οι Σουηδοί. Οι Σουηδοί έχουν τόσο μεγάλο ενεργειακό δυναμικό onshore Εκεί έχουν πολλέ ε, κρυφέ ατζέντε νομίζω οι Σουηδοί και δεν έπαιξε καθαρό παιχνίδι η Σουηδική κυβέρνηση διότι μάλιστα πρόκειται και για ένα έργο που είχε πάρει και χρηματοδότηση από το Recovery Plan. Για το τρίτο, για την εναρμόνιση, είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει με λεπτομέρεια. Το μέγα πρόβλημα που βλέπω είναι η εναρμόνιση των διαμεθοριακών δομών. Πρόσφατα συζήτησα με μια δανέζικη επιχείρηση που είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στην Βόρεια Θάλασσα είναι οι Δανείοι, είναι οι κατοχώρες, είναι οι Εγγλέζοι, μου είπαν καθαρά ότι τα support scheme δεν είναι πρόβλημα. Εάν θα γίνει με πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος στη Δανία ή με άλλο σύστημα στην Ολλανδία, αυτό δεν είναι για αυτούς το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι, για παράδειγμα, ο αγωγός από Δανία σε Ενωμένο Βασίλειο συζητιέται τώρα ανάμεσα στα εθνικά δηλαδή στο National Grid το αγγλικό και στο αντίστοιχο δανέζικο. Το ζήτημα είναι πόσο γρήγορα θα υπάρξει αυτή η διασύνδεση γιατί από την ε, Ανατολική ε, ακτή της Αγγλίας εκεί είναι και θέματα ανέμων τέλος πάντων ε, εγώ για τους ρυθμιστές βλέπω το πράγμα το ίδιο. Το πρόβλημα των ρυθμιστών και η νοοτροπία τους. Γιατί εμείς τους βάλαμε για να μειωθούν τα μονοπόλια στα δίκτυα. Να μειωθεί το κόστος για τον καταναλωτή. Γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκαν. Και τώρα μπαίνουμε σε μια νέα εποχή και αυτή η νέα εποχή δεν είναι μονάχα η νέα εποχή των εναλλακτικών ενεργειών. Είναι και της ε, ολοκλήρωσης των δικτύων και υπηρετικά Μάλιστα σε ορισμένε χώρες έχουμε πολύ παλαιά δίκτυα που πρέπει να εξυγχρονιστούν και πρέπει να βρεθεί ένα modus συμβέντη με τους ρυθμιστέ. Θα διαβάσω προσεκτικά και αυτό το θέμα με τον κεφαλογικό εξοπλισμό. Με τον εξοπλισμό με κεφάλαια μάλλον. Εκεί βρίσκεται και η διασύνδεση με, τα, με τους νέους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. Τώρα, εγκρίσεις νέων υποδομών. Αυτό είναι πολύ καυτό θέμα και για μας τους πράσινους. Ε, προσπαθούμε να είμαστε πολύ υπεύθυνοι στην προσέγγισή μας. Μου λέγουν πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο για καλωδιακές ε, διασυνδέσεις. Είναι ευχάριστο που υπάρχουν και νέες εφαρμογές, για παράδειγμα, ε, τεχνολογικές και υπάρχουν και νέες είναι άνθρακα. Υπάρχουν τώρα ε, καλώδια, ε, ε, είναι που μπορούν να μεταφέρουν πολύ μεγάλη ποσότητα ηλεκτρισμού και μπορώ να παραμείνω στην ίδια γραμμή διότι οι μονοτήρες βιδώνονται πάνω στην ίδια την αγωγή, στην ίδιο τον αγωγό, ενώ λόγω ανέμων πρέπει στις, ε, στους πυλώνες, τους παραδοσιακούς πυλώνες να υπάρχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των μονοτήρων. Είναι τέλο πάντων τεχνολογικές εξελίξεις που είναι ενδιαφέρον να τις παρακολουθήσουμε. Σε αυτό το θέμα της καινοτομίας πρέπει να προβλέψουμε και ένα συγκεκριμένο χρηματοδοτικό μηχανισμό Μιλούμε για παγκόσμιες εταιρείες τώρα. ABB, Alstom και Siemens. και ο πρώην ε, ε, ε, Ιταλός κατασκευαστής ελαστικών. Μιλούμε για τεράστιες επιχειρήσεις. Τώρα μπαίνουν και οι μεγάλες επιχειρήσεις ε, software οι αμερικανικές μπαίνουν και οι Κινέζοι. Έχουμε λοιπόν ειδικά στο θέμα αυτό των υποδομών ανάγκη να δημιουργήσουμε ένα νέο χρηματοδοτικό μηχανισμό. Ένα ερώτημα τώρα. Merchant Lines. Πώς το βλέπετε αυτό. Υπάρχει αυτή η Merchant Line μεταξύ Ενωμένου Βασιλείου και κάτω χωρών. βλέπετε να μπορέσει να ε, εξελιχθεί το δίκτυο αυτό και μέσω ε, merchant lines. Το ερώτημα που τίθεται ακόμα για μένα είναι αυτό το μνημόνιο συμφωνίας που αναφέρατε. Μου φαίνεται ενδιαφέρον. Εκεί που ανησυχούν οι επενδυτές αλλά και αυτοί που έχουν τα δίκτυα είναι πώς μπορεί να συζητηθεί το πράγμα αυτό αλλά ταυτόχρονα τα έργα που πρέπει να επιταχυνθούν, να προχωρήσουν γρήγορα δηλαδή, να μην παρεμποδιστούν. Ευχαριστώ και εγώ από πλευρά μου για τα σταρά τα λόγια σας. Γνωριζόμαστε εδώ και καιρό και εγώ σας ξέρω ότι δεν μασάτε τα λόγια σα και από άλλη ε, δραστηριότητα που είχατε στο παρελθόν. Και σήμερα το πρωί συζητήσαμε για τις υποδομές και εδώ έχουμε καταλάβει και εμείς και πρέπει ε, να προχωρήσουμε στα θέματα των ρυθμιστικών αρχών. Εμείς επιβάλαμε αυτές τις δομές για τον ανταγωνισμό, αλλά δεν θα πρέπει αυτό να στραγγαλίζει την οικονομική δραστηριότητα. Κάτι άλλο τώρα. Ε, συζητάμε αν θα είναι εναέριες ή υπόγειες οι συνδέσεις στα καλώδια. Εγώ είμαι από το Βερολίνο και στα βόρεια του Βερολίνου είναι προστατευόμενη φυσική ε, περιοχή Δρυμός ε, και τίθεται το θέμα αν θα είναι αέρια τα καλώδια ή θαμμένα. Ε, για να θάψει ένα καλώδιο είναι πολύ ακριβό όμω, και δεν είναι μόνο το κόστος αλλά ε, τι θα γίνει ε, και με τη γραμμή την ίδια. Δεν θα πρέπει από πάνω η φύση να αφαιθεί να ξανέρθει σε άγρια κατάσταση επειδή είναι προστατευόμενη περιοχή. Κάτι άλλο που θα ήθελα να σας ρωτήσω από την εμπειρία σας, το συζητήσαμε και εδώ και χτες σε πιο περιορισμένο κύκλο. Όταν έχουμε προγράμματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και τα οποία χαρακτηρίζουμε ως τέτοια και τα προβάλλουμε επί τόπου, ένα σημείο διασύνδεσης ή κάτι τέτοιο, Και μήπως ε, πέσουμε στην παγίδα που έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι, γιατί ο κόσμος που έχει επιτόπου προβλήματα και ε, διαμαρτύρεται και αντιστέκεται και δεν το θέλει, έχουν και την Ευρώπη πλέον ως αποδιοπομπαίο τράγο, α, ότι η Ευρώπη το θέλει το πρόγραμμα και ε, αντιδρούν ακόμα περισσότερο. Αυτό πώς μπορούμε να το αποφύγουμε. Αυτά, ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Πρόεδρε, σήμερα το πρωί συζητήθηκε σύντομα ε, η υποδομή ε, για το 2020 και μετά. Είναι σημαντικό θέμα αυτό και έχουμε εργαστεί και από πλευρά Κοινοβουλίου για τι επιλογές για τα αεολικά πάρκα ε, στην ανοιχτή θάλασσα και το recovery plan που είπατε κι εσείς για το ε, θέμα της χρηματοδότησης από το σχέδιο ανασυγκρότησης. Αλλά ε, είναι τόσο διαφορετικά τα εθνικά προγράμματα και τα έργα που υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσει Στην Ολλανδία, παρόλο που έχουμε πολύ μεγάλες υποδομές ε, και έχουμε πολύ μεγάλες νομοθετικές παρεμβάσεις με μεγάλες αλλαγές στους νόμους ακριβώς αυτά τα έργα τώρα εσείς πώς μπορείτε να τα συνδέσετε και με την νομοθεσία πολύ καλή ιδέα να κατονομάσουμε κάποια προγράμματα και να τα χαρακτηρίσουμε διασυνοριακά, ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος κτλ. Δεν θα πρέπει μόνο να εμβαθύνουμε, αλλά να τα συνδέσουμε και με την νομοθεσία. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτά και θέλω να τονίσω ότι θα διαβάσω με μεγάλο ενδιαφέρον την έκθεσή σας και το είπε και ο κύριος Τούρμες ότι πολύ σύντομα θα πρέπει να έχουμε κάποιες διασυνδέσεις. Δεν μπορεί ο κόσμος να επενδύει και να φτάνει σε στόχους αν δεν έχει τις βέλτιστες δυνατές διασυνδέσεις. Ευχαριστώ. Καλώς. Η συνάδελφος Χολ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε για το, για την σημαία, για το κρίκες φλακ. Κυρίως ε, θα ήθελα να ε, μου πείτε ποια θεωρείτε, ποιες θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι οι συμβατικές υποχρεώσεις οι οποίες ε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη γιατί διαφορετικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθει κανείς σε συμφωνία για τα offshore grids. Νομίζω ότι και άλλωστε πρώτη φορά γίνεται αυτό στο παρελθόν δεν αντιμετωπίσαμε με τον ίδιο τρόπο τα προβλήματα αυτά. Κύριε Ντάμοβιτς, έχετε το λόγο. Και να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις με χρήβη 100% και σύντομα. Ευχαριστώ για το πακέτο το οποίο με φορτώσατε. Ευχαριστώ κύριε Τούρμερς, το έχουμε ξανασυζητήσει. Ε, δεν διαφωνούμε. Ε, ξέρω για τη δική σας πολιτική ομάδα, αλλά και για άλλες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για το θέμα των εμποδίων για την αδειοδότηση. Ε, το θέμα για τη χλωρίδα, την πανίδα και ε, την προστασία της φύσης το καταλαβαίνω. Καμιά φορά όταν συζητούμε για τους στόχους, τους αηφόρους και τις υποδομές που απαιτούνται προσκρούμε σε άλλα προβλήματα. Και μένα ε, με αυτό όταν βλέπω κάποιο συγκεκριμένο έργο. Ε, τι να κάνουμε, 100% δεν μπορεί να υπάρξει λύση και είναι σημαντικό η Ευρώπη να το συζητάει. Και έχουμε διαφοροποιημένες στρατηγικές ε, αηφορίες. Από τη μια θέλουμε να έχουμε φύση και από την άλλη ενέργεια. Πώς θα τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο γιατί έχουμε και αντικρουόμενους στόχους καμιά φορά. Ε, σιγά σιγά πρέπει να αρχίσει να μας απασχολεί αυτό και με κάποια ειλικρίνεια και τιμιότητα απέναντι στην κοινωνία των πολιτών. Γιατί έχει απέτηση, έχει αξίωση από την πολιτική ο κόσμος να ασχολείται και με αυτά τα θέματα, τη σύγκρουση των στόχων μας. Ε, πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα, για όλα αυτά τα θέματα, τα τεχνικά προβλήματα που αναφέρεται, και για την οικονομία. Ε, μεγάλη ευκαιρία για την Ευρώπη, συμφωνώ. Συζητήστε το και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάπου πρέπει να γίνει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι εθνικές λογικές και να υπάρξει μια άλλη νοοτροπία ε, υπέρ των ευρωπαϊκών πιλωτικών ε, προγραμμάτων και έργων. Γιατί πρόκειται για τριψήφια εκατομμύρια. Εκεί τα νούμερα, αυτή είναι η τάξη μεγέθους. Και ε, μόνο συντονίσουμε τις δυνάμεις μας. Ε, τώρα, για, κύριε Τούρμας, αυτό που είπατε για τη γραμμή ε, Ηνωμένου Βασιλείου Ολλανδίας, εντάξει δεν έχω κανένα πρόβλημα με τη σύνδεση, αλλά να το απαντήσω διαφορετικά. Το είπα και στην εισαγωγική μου ομιλία. Είμαι ακράδαντα πεπισμένος ότι το θέμα της ενιαίας ε, ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι κάτι το οποίο θα παίξει ρόλο να, να, να, γίνει πραγματικότητα πέρα από τα χρηματιστήρια και τις τιμές. Θα πρέπει να βρούμε ένα κοινό ορισμό ε, για ε, τη σκοπιμότητα μιας τέτοιας ε, αγοράς και όλα τα υπόλοιπα λύνονται και το θέμα Ηνωμένου Βασιλείου ε, ένας ε, κανονικός επενδυτής ε, που φτιάχνει μια γραμμή, που την κατασκευάζει, δεν μπορεί να έχει απέναντί του τρει-τέσσερι αγορέ, τρει-τέσσερι μηχανισμού και ρυθμιστικέ αρχέ. Δεν έχει νόημα να την κάνει την επένδυση. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Από την άλλη, όταν μιλάμε για μια ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική και θέλουμε να την υποστηλώσουμε και ε, με μια σωστή αγορά σε πλαίσια αγωνισμού για να λειτουργεί, αλλιώς δεν λειτουργεί, τότε ε, χρειάζονται ευρωπαϊκά κριτήρια ε, και πρέπει να τα συζητήσουμε για μια ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρώπη, μια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και πώς θα λειτουργεί. Δεν γίνεται αυτή η συζήτηση. Η συζήτηση γίνεται στο οικονομικό πλαίσιο, όχι της ενέργειας. Μόνο έτσι ε, θα μπορούμε να βρούμε και τα οικονομικά για τη δημιουργία των δικτύων. Έτσι απαντώ αυθόρμητα ε, στα όσα είπατε εσείς. Κύριε Γκλάντε, το θέμα των, ε, της εναέριας γραμμής του καλωδίου του υπογείου ε, ε, Διαβάστε το έγγραφο που συζήτησε και συνεννοήθηκε και κατέληξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τους κατασκευαστές καλωδίων στην Ευρώπη. Το κάθε ε, έργο έχει την ιδιαιτερότητά του. Δεν μπορούμε να πούμε πάντα ότι είναι καλό το καλώδιο και κακή η εναέρια γραμμή. Αλλά κοιτάξτε, μιλήσαμε τώρα για τα θέματα της προστατευόμενους δρυμούς για να βάλετε 700 ε, μέτρα ε, καλωδίου ε, είναι 26 τόνους το καρούλι και χρειάζεστε μια ταλίκα 30 τόνων για να μεταφέρετε 26 τόνους καρούλι. Εγώ Έχω ζήσει στην Ευρώπη και δραματικές συζητήσεις ε, και είμαι και ακρεφνής Ευρωπαίος. Αυτό που μου λέτε επί τόπου το έχω ζήσει. Γιατί ε, όταν του ζήσει είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα, σου λέει Α, θα έρθουν οι Ευρωπαίοι τώρα από τι Βρυξέλλε να μα πούνε και πού θα βάλουμε τα καλώδια μα για το ρεύμα είναι προγράμματα των Εθνικών Κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής και του Κοινοβουλίου και σκεφτήκαμε να γίνει διασυνοριακή σύνδεση και θα πρέπει να τους πείσουμε ότι δεν είναι καμιά εφεύρεση των Βρυξελών που ήρθε εδώ να ε, ταλαιπωρεί τους ανθρώπους ε, εκεί που ζουνε. Γιατί βγαίνει και ένας ευρωπαϊκός σοβινισμός που καμιά φορά μας τρομάζει αλλά και εδώ δεν μασάω τα λόγια μου. Και θα είχα μια συμβουλή να δώσω. Και για το άρθρο 194 ε, της συνθήκης. Δεν είναι κάτι που εφήβρε ε, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε το Κοινοβούλιο. Είναι μια διαδικασία ετών για το πού ε, ε, είναι στην Ευρώπη οι αρμοδιότητες και πώς καταλήξαμε στην ευρωπαϊκή αυτή συνθήκη. Και αυτό θα πρέπει να το εξηγήσουμε στον κόσμο για να κερδίσουμε ε, τους ανθρώπους ότι έχουν συμφωνήσει και τα κοινοβούλια και οι κυβερνήσεις. Αλλιώς δεν θα είχε προκύψει ποτέ το άρθρο 194. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη ευρωπαϊκή πώς το... διαπαιδαγώγηση ότι ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούν από μόνα τους να τα αποφασίζουν αυτά, αλλά ε, και οι κυβερνήσεις πρέπει να εξηγούν την Ευρώπη και τα προγράμματα υποδομών που είναι υπέρ της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Συμφέροντος. Χρειάζεται πολύ δουλειά εδώ. Και μια που έχω το λόγο και κάνω και διαφήμιση για τον εαυτό, του, εαυτό μου, ε, Έκανα και πέρυσι μια έκθεση για το ε, Salzburg και ασχολήθηκα πάρα πολύ με το πώς συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών. Έκανα συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες συζητούνται τώρα επιθετικά με αντιπαράθεση ε, στο Salzburg, Ότι τι ρόλο μπορεί να παίξει ένα κοινοβούλιο, εθνικό ή περιφερειακό, ε, στις αποφάσεις για ένα έργο και πώς μπορεί να είναι ο υπερασπιστής των συμφερόντων των πολιτών. του. Δηλαδή όλα αυτά δεν χρειάζεται να τα εφεύρουμε από την αρχή αλλά να εξηγούμε στον κόσμο τι συμβαίνει. Και τι συμβαίνει στο Σάλτσμπουργκ. Ε, ε, ε υπήρξε μια ολόκληρη προσπάθεια, κόπος, αγωνία 10 ετών και οδήγησε σε πολύ έντονες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις. Αλλά το συζητούμε με τις ε, πρωτοβουλίες των πολιτών, ο Δήμαρχος, με, τη ε, με την τοπική βουλή, κυβέρνηση κτλ. Οι εταιρείε. Κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί αυτός ο διάλογος και ε, πιστεύω ότι η διαδικασία από και πέρα μπορεί να είναι απλή. Θα βρείτε στην έκθεσή μου και μια έκθεση... Ε, πεπραγμένων. Ε, ε, τι έχει κάνει η Αυστρία, ας για την εφαρμογή των όσων ε, εγώ προτείνω και το πρόγραμμα 380. Κιλοβόλτ. Και πολιτικά να τα εξηγούμε όλα αυτά στον κόσμο. Επαναλαμβάνω, δεν πρέπει κάθε φορά να ε, εφευρίσκουμε τον, τον τροχό, αλλά να εξηγούμε στον κόσμο τι συμβαίνει και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κύριε Ρόι πώς σας είπα. Α, Ρόι Α, ε, ε, είστε συγγενείς του ποδοσφαιριστού. Ε, όχι, όχι, εγώ δεν είμαι επιθετικός, είμαι μάλλον μέσος, είμαι λιγότερο καλός. Καλά, ε, βγάζουν και πιο πολλά λεφτά αυτοί από εσά. Έχουμε τώρα το εξή πρόβλημα. Έχουμε πολλά εθνικά προγράμματα συνδέσεων με ολικά πάρκα στη θάλασσα αλλά ε, χρειάζεται τώρα και ένα δίκτυο που να συνεχίζεται στην ενδοχώρα και στη Βόρεια Θάλασσα και στη Βαλτική. Γι' αυτό έγινε αυτή η προσπάθεια στη Βόρεια Θάλασσα των 10 χωρών που βρέχονται από τη θάλασσα αυτή. Ε, εντάξει, κινητοποιούνται και οι επενδύσεις, αλλά το θέμα από εκεί πέρα γίνεται εθνικό γιατί το ρεύμα που παράγεται μπαίνει στα εθνικά δίκτυα. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα μοντέλο για ένα ευρωπαϊκό δίκτυο και για ένα άλλο λόγο. Το είπα και προηγουμένω. Έχουμε τεράστιο δυναμικό στη Βόρεια Θάλασσα και στη Βαλτική. Εντάξει. Αλλά έχουμε το πρόβλημα της ισορροπίας δυνάμεων. Τι γίνεται όταν έχω ένα πελάτη κάπου στην Ευρώπη που χρειάζεται ρεύμα και δεν φυσάει. Δηλαδή θα πρέπει κάπως να εξισορροπούμε ε, την άπνοια με άλλα υδροελεκτρικά εργοστάσια, κάτι τέτοιο που να πηγαίνει το ρεύμα είναι δεδομένο ότι θα έχει καταναλωτήσει πάντα ρεύμα και με άπνοια. Και έρχομαι στο Kriegers Frag τώρα και αυτά που ρώτησε η κυρία Χολ. Στα ε, προγράμματα που έχουμε θα πρέπει να κοιτάμε πώς μπορούν στη συνέχεια να γίνουν τεχνικές ε, προσαρμογές για να γίνει ευρωπαϊκό το δίκτυο. Εξού και η Γερμανία και η Δανία συνεχίζουν τις προσπάθειες για τους επενδυτές και τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας. Δεν το λέω τεχνικά τώρα, αλλά στο Kriegers Flag μένουν ανοιχτές τώρα οι διασυνδέσεις όταν δεν ήσουν οι ε, Σουηδοί να επιστρέψουν να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Είναι ευρωπαϊκή η ανάγκη και τεχνικά και πολιτικά και για τη ρύθμιση και για ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Αντάμοβιτς. Äh, äh, Πραγματικά έχετε έναν τρόπο να τα λέτε με τόση ακρίβεια και τα πράγματα με το όνομά τους ε, πολύ θετικό, θα μας βοηθήσει σίγουρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Καλή δύναμη. Είμαι βέβαιος ότι θα σας ξαναδούμε σε διάφορα φόρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς για την υπέρβαση ωραρίου. Λήξη συνεδρίασης.